Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, ήρθατε στην ε, κοινή συζήτηση για το σύστημα εισόδων-εξόδων για την καταγραφή δεδομένων εισόδων-εξόδων καθώς και άρνηση εισόδου υπηκών τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς επιβολής του νόμου. Και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί. Έχουμε δε προσκαλέσει εκπροσώπου τη ευρωπαϊκή επιτροπή, καθώς και του οργανισμού EU-LISA. Καλώ ορίσατε. Η e EU-LISA είναι αρμόδια, ο οργανισμό δηλαδή είναι αρμόδιος για τις τεχνικές ε, λεπτομέρειες. Έχουμε λάβει ως τώρα μια έκθεση του λίσα σύμφωνα με, τον με το άρθρο του κανονισμού, και η έκθεση είναι διαθέσιμη στα έγγραφα συνεδριάσεως. Ας δώσουμε το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στους συναδέλφους ε, του Ιγιουλίσσα για να προχωρήσουν σε παρουσίαση για 15-20 λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους μας, την κυρία Γκάλ, και, δηλαδή, και τον κύριο Δίας Τεμέρα, όταν θα ε, προσέλθει. Ας αρχίσουμε την συζήτηση με την πρώτη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορίστε παρακαλώ ο Ευχαριστώ και καλημέρα. Από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών για τα project εφιών συνόρων που περιλαμβάνει και το σύστημα αιτιός, αιτία συγγνώμη, εξόδων εισόδων. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε στην πρώτη αυτή συζήτηση για την εφαρμογή των συστημάτων και για την ε, πρόοδο των εργασιών. Η προπαρασκευή των δύο συστημάτων προχωρεί καλά σε συνεργασία με τις χώρες μέλη και τους διαφόρους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Ως ίσως γνωρίζετε, το σύστημα αποτελείται, μάλλον βασίζεται σε διαφορετικά νομοθετικά κείμενα. Οι διατάξεις του κανονισμού ΕΤΙΑΣ προβλέπουν ότι τα δύο συστήματα θα λειτουργούν εκ θα, θα συνεργάζονται. Για το σύστημα εισόδων-εξόδων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδρύσει σχετική επιτροπή όπου συζητούνται τα θέματα αυτά με, τις, με τους εκπροσώπους των χωρών μελών. Πρώτη σειρά εκτελεστικών μάλλον πράξεων, 10 δηλαδή κείμενα συνολικά, βιομετρικά, login, data management, η συνεργασία μεταξύ των δύο συστημάτων, θεωρήθηκαν ως προϋποθέσεις για την αρχή της εφαρμογής του συστήματος εισόδων-εξόδων. Γίνεται συνεργασία με τον Ιουλίσα και συζητούνται στην Επιτροπή που προανέφερα με τους εκπροσώπους των χωρών μελών. Τα κείμενα έχουν εγκριθεί στην Επιτροπή αυτή και έχουν περάσει από δημόσια διαβούλευση μέσω μηχανισμού feedback. Έχουν περάσει τις εσωτερικέ διαδικασίες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ευθυγραμμιστεί και με τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτου Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, ώστε τα κείμενα να είναι πλήρως προετοιμασμένα, προσαρμοσμένα και έτοιμα μέσα Φεβρουαρίου. Επειδή τα κείμενα αυτά και ιδίως τα τεχνικά τους στοιχεία θεωρούνται σταθερά σε συμφωνία με τις χώρες μέλη και με τον οργανισμό EU που έχει αναλάβει το τεχνικό μέρος τα τεχνικά αυτά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχέδια των ε, εφαρμοστικών διατάξεων έχουν ενταχθεί στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί για την εφαρμογή του συστήματος. Τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού έχουν υποβληθεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκδώσει αυτή επίσημη γνωμοδότηση, η διαδικασία η οποία συνεχίζεται και η επίσημη γνωμοδότηση της Επιτροπής θα είναι έτοιμη στα, στη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Εκτός από αυτές τις ε, εκτελεστικές πράξεις, που είναι σχεδόν εγκεκριμένε, έχουμε τέσσερις πράξεις ακόμα στην προπαρασκευαστική φάση, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για να αρχίσει η τεχνική εφαρμογή του σχεδίου, αλλά θα πρέπει να εγκριθούν πριν από την αρχή της εφαρμογής του συστήματος. Τέσσερις λοιπόν implementing acts που παραμένουν και ε, αναφέρονται στο σύστημα που θα χρησιμοποιούν οι φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων καθώς και μια διαδικασία fallback, ιστοσελίδες με γενικές πληροφορίες για το κοινό σχετικά με το σύστημα εισόδων-εξόδων και πληροφορίες για την διάβαση μεθορίων και ένα έγγραφο template για πληροφορίες για το κοινό πού θα είναι διαθέσιμο το κείμενο αυτό στις διαβάσεις των συνόρων. Για το web service κυρίως που θα χρησιμοποιούν οι φορείς, επειδή υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις στον κανονισμό αιτίας και υπάρχουν και πρόσθετες διατάξεις οι οποίες αναφέρουν ότι η διαβούλευση με τους ε, φορείς carriers ε, θα πρέπει να γίνουν πριν από την έγκριση του κειμένου, έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύσεις με τους carriers και προχωρεί έτσι ώστε να καθορίσει τους τρόπους εφαρμογής του, της διαδικτυακής αυτής υπηρεσίας, web service. Από την ε, οπτική γωνία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι τεχνικές προπαρασκευές για την εφαρμογή του συστήματος πηγαίνουν καλά. Η καταληκτική ημερομηνία που έχουν συνυπογράψει τα διάφορα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή του συστήματος θα γίνει σεβαστή και εκ με την προπαρασκευαστική αυτή εργασία έχουμε αρχίσει και την προπαρασκευή για τη σύνταξη εγχειριδίου που να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει κοινή βάση για τους χρήστες του συστήματος, κυρίως δηλαδή τερανοφύλακες της διαβάσης των συνόρων. Αυτό γίνεται πάλι σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Για τις χώρες μέλη τώρα έχει αρχίσει η προπαρασκευή πρώτα για τις διασυνδέσεις τους με το σύστημα, ότι θα πρέπει δηλαδή να διασυνδέσουν την υποδομή ε, προστασία των συνόρων και τα ηλεκτρονικά του συστήματα με το κεντρικό σύστημα του συστήματος ΕΕΣ. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια τώρα για όλε τι χώρε μέλη. Εκ παραλίλου οι χώρε μέλη έχουν αρχίσει επίση να εργάζονται για την προετοιμασία των σημείων διαβάσεων των συνόρων με τη χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη χρήση του συστήματο και ιδίω βιομετρικών συσκευών που θα επιτρέπουν την καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως απαιτεί ο κανονισμός, αλλά και κάμερες που θα μπορούν να λαμβάνουν ε, φωτογραφίες του ταξιδιώτη, πάλι όπως απαιτεί ο κανονισμός. Τέλος, οι χώρες μέλη έχουν αρχίσει να σκέπτονται την αυτοματοποίηση των διαβάσεων των συνόρων. Αυτή η δυνατότητα θα ανοιχθεί μέσω, μέσω τροπολογιών του κώδικα Schengen που έχουν εγκριθεί εκ παραλλήλου με, που θα εγκριθούν μάλλον με, με την έγκριση του συστήματος εισόδων-εξόδων. Σε ό,τι αφορά το σύστημα αίτιας, ως γνωρίζετε, αυτό το σύστημα εγκρίθηκε μόλις προ λίγων μηνών και έχουμε μακρότατο κατάλογο πράξεων, κατεξουσιοδότησης και εκτελεστικών που πρέπει να εγκριθούν. Ο συνολικός του αριθμός είναι 21 εκτελεστικές πράξεις και 14 κατεξουσιοδότηση. Από αυτές θεωρήθηκε ότι 12 εκτελεστικές και 3 κατεξουσιοδότηση είναι αναγκαίες για να αρχίσει η τεχνική εφαρμογή του, συστήματος, του κεντρικού συστήματος αιτιάς σε συμφωνία με τις χώρες μέλη και με τις εργασίες των ομάδων εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια έχουμε ήδη συμφωνήσει με τις χώρες μέλη, τους εμπειρογνώμονες χώρων μελών για τις τρεις ε, εκτελεστικές πράξεις που πρέπει να εγκριθούν ταχύτατα, τρεις επίσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες αφορούν υπηρεσίες που θα χρησιμοποιούν οι ετούντες για να λαμβάνουν περισσότερες προφορίες, ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει στον ετούντα να πληροφορηθεί την πρόοδο της αιτήσεώς του, και τέλος ένα εργαλείο για ετούντες ή μάλλον αυτούς που ήδη κατέχουν άδεια ταξιδίου για να μπορέσει να ζητήσει τη διατήρηση των δεδομένων στο σύστημα. Προχωρούμε επίσης για 7 από τις 12 εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να αρχίσει η εφαρμογή του αιτίας. συνεχίζεται η εργασία για την διαχείριση δεδομένων και επίσης για σημεία πρόσβασης για τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, για την συλλογή των προσωπικών δεδομένων μέσω των εντύπων αιτήσεων. Αναμένουμε να ολοκληρώσουμε το έργο για τις 12 ε, αυτές εκτελεστικές αποφάσεις ε, ως το δυνατόν συντομότερο, μέχρι τέλους Φεβρουαρίου φέτος δηλαδή, ώστε να επιτρέψουμε στον Ιουλίσα e να αρχίσει το δυνατόν συντομότερο την τεχνική εφαρμογή του συστήματος και πρώτα-πρώτα με την κατάστρωση των τεχνικών προδιαγραφών που είναι αναγκαίες για να εφαρμοστεί το σύστημα. Εκ παραλλήλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει όπως τη ζητήθηκε από το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού αιτιάς έχει συντάξει και διαδοχικές τροπολογίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του ΕΤΙΑΣ, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές μάλλον τροπολογίες, που απορρέουν από το ότι ο ΕΤΙΑΣ θα αντικαταστήσει άλλα συστήματα Αυτές οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί στις 7 Ιανουαρίου φέτος. Σε ό,τι αφορά την προπαρασκευή της εφαρμογής του αιτιάς, η διαδικασία είναι περίπλοκη, με εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων φορέων, πρώτα-πρώτα τρεις διαφορετικοί οργανισμοί που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του project. Επίσης, στο επίπεδο των χωρών μελών είναι διαφορετικές οι αρχές οι οποίες θα πρέπει να εμπλακούν στην διαδικασία αξιολόγησης της ε, αίτησης άδεια ή της έγκρισης άδεια, της έγκρισης ε, ταξιδιού μάλλον, Τώρα, για την εφαρμογή θα πρέπει πρώτα να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Δεύτερο, συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αρχών που θα πρέπει να συνεργάζονται για να, για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την άδεια ταξιδιού ενώ η συνεργασία αυτή δεν είναι δεδομένη πάντοτε. Άρα χρειάζονται πολλές τροποποιήσεις και να υπάρξει σημαντική πρόοδος στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι διάφορες αρχές, στο εθνικό επίπεδο κυρίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει ένα γύρο των πρωτευουσών, ώστε να προκαλέσει πρόοδο στην ε, διαδικασία αυτή και για να προχωρήσει και μέσα στον χρόνο η εφαρμογή του συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σιλόν. Όπως είπατε, ο Ιουλής έχει αναλάβει αυτό το σημαντικό και περίπλοκο καθήκον. Θα ακούσουμε από τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συστήματος Εσόδων-Εξόδων, κύριο Συρίγο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο καθήκον ο Ιουλίσσα. Ε, έχετε το λόγο σας παρακαλώ, λάβετε, ε, ανοίξτε το μικρόφωνο. Good morning. Ε, my name is Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φάνη Σιρίου, ονομάζομαι και είμαι ο Πρόεδρος ε, αυτής της συμβουλευτικής ομάδας για το σύστημα εσόδου-εξόδου και όσον αφορά τις άλλες ε, λειτουργίες και σχέσεις του συστήματος. Να σας πω τι κάνουμε και για τα δύο συστήματα. Σύμφωνα το σύστημα εισόδου-εξόδου, ξεκινήσαμε μια προπαρασκευαστική εκστρατεία όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος, παράλληλα και με τη διαδικασία της έγκριση της νομικής βάσης. Έτσι θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια εύρεθμη λειτουργία του συστήματος. Μόλις υπάρξει η νομική βάση Θεωρούμε ότι είναι σωστή αυτή η προσέγγιση και έτσι νομίζουμε ότι η υπηρεσία πρόκειται να επιτελέσει διάφορες λειτουργίες και όσον αφορά την προετοιμασία των ε, διαγωνισμών, των προμηθειών, την ε, συγκεκριμενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σιλών, δηλαδή το πώς θα υπάρξει στενή συνεργασία με την Επιτροπή για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τις σχεστικές εφαρμοστικές πράξεις. Οπότε ετοιμάσαμε αυτή, ε, τον διαγωνισμό για τις ε, προμήθειες και στη δημόσια σύμβαση τέλος πάντων έγινε η α, ε, κλίση για υποβολή ενδιαφέροντας τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και όσα πρότεινε και επίσης έχουμε ετοιμάσει την ενδελεχή ε, ενδεικτική ε, διαδικασία προγραμματισμού για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα σε εθνικό επίπεδο, σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την ε, εποπτεία των εποπτικών φορέων. Το Advisory Group, το Διοικητικό Συμβούλιο μας και λοιπά. Ο αρχικός προγραμματισμός για την ε, εφαρμογή ε, πέστη τις τελευταίες πινελιές, αλλά ακόμα επεξεργαζόμαστε το τι θα γίνει στην ε, ομάδα των συμβούλων, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες, τις διάφορες ροές λειτουργίας. Ε, θέλουμε να καταλάβουν όλοι περί τίνος πρόκειται και έτσι να προετοιμαστούν ακριβώς όπως προβλέπει αυτός ο προγραμματισμός που θα έχει ολοκληρωθεί μόλις έχουμε ολοκληρώσει τις συμβατικές ε, ε, ρυθμίσεις και έτσι θα προχωρήσουμε κατά το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή αρχάς Απριλίου. Αυτές οι εφαρμοστικές ε, λειτουργίες, λειτουργίες υλοποίησης θα έχουν να την προετοιμασία του συστήματος το εθνικό Interface που το ονομάζουμε ΝΟΥΙ από τα αρχικά του, ε, τις υπηρεσίες ε, δικτύου, τις, ε, τα θέματα επικοινωνιών, το βιομετρικό σύστημα, τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν στο σήμερα ισχύον VIS και το σύστημα που συντεριάζει τα βιομετρικά στοιχεία και επίσης το κεντρικό μητρό αρχείο όσον αφορά τις αναφορές στατιστικών στοιχείων. Η πρόοδος ε, αυτής της εργασίας παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι θα ξεκινήσουμε την διαδρομή αυτή της υλοποίησης των 36 μηνών η οποία ξεκίνησε ήδη από πέρσι. Τώρα κάποια πρακτικά στοιχεία όσον αφορά την υλοποίηση του συστήματος εισόδου-εξόδου. Έχουμε τρεις ε, άξονες ε, που αφορούν τις ε, τεχνικές προδιαγραφές, τον διαγωνισμό αλλά και την προετοιμασία. Ακριβώς όπως είπατε και στην αρχή, Πρόεδρε, που είναι ο πρώτος άξονας, η υποβολή των εκθέσεων. Θα πάμε τώρα για τη δεύτερη έκθεση που τώρα είναι στη διαδικασία της σύνταξης και την οποία θα λάβετε την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Και έτσι θα μπορέσετε να έχετε ε, μια σφαιρική άποψη για τη δουλειά μας. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα των ε, προσλήψεων. Έχουμε προσλάβει 14 ε, υπαλλήλους προσωρινούς τρεις για οικονομικά και 11 για τεχνικά θέματα και επομένως αυτό είναι το νέο μας προσωπικό και αυτοί έχουν ε, πάρει τις θέσεις τους και έχουν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο πέρσι. ο πλευρά τώρα του διαγωνισμού, όπως είπαμε προηγουμένως, ήδη έχουμε αρχίσει τη δουλειά από το τρίτο τρίμηνο του 16 και τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει ούτως ώστε να καταλήξουμε σε ένα σωστό σύστημα. Οπότε, έχουμε χωρίσει σε δύο τη δουλειά μας. Πρώτα-πρώτα, λεπτομέρειες για το ίδιο το κεντρικό σύστημα. Και, κατά δεύτερον, έχουμε τις λεπτομέρειες, τα στοιχεία για το σύστημα που συντεριάζει, που ταυτοποιεί τα βιομετρικά στοιχεία. Και συμπεριλαμβάνονται εδώ και οι προδιαγραφές για το Workflow Engine. Είναι τεχνικό θέμα, μια τεχνική λύση που μας οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την δουλειά μας στα σύνορα. Τώρα, όσον αφορά αυτόν τον διαγωνισμό, έχουμε την πρώτη φάση που έχει ξεκινήσει όσον αφορά τον διαγωνισμό. Αυτό ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και ήδη έχουμε λάβει τις απαντήσεις, τις προσφορές Γίνεται τώρα η αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 18. Δεύτερη φάση ξεκίνησε αρχάς Οκτωβρίου του 18, 9 δεκάτου συγκεκριμένα και συμπεριλαμβάνονται και τα θέματα των προδιαγραφών που σας είπα προηγουμένως, η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών ε, ήταν για αρχάς Ιανουαρίου, 3, 3 Ιανουαρίου φέτος και στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι γίνεται η αξιολόγηση τώρα και τελικά θα γίνει η υπογραφή του βασικού, του, του, του, συμβάσεως πλαισίου κάποια στιγμή κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου ή αρχάς τέλος πάντων Απριλίου φέτος. Τώρα, για το διαγωνισμό που αφορά το BMS και τις προμήθειες μας στην πρώτη φάση αυτής της ε, διαδικασίας της ε, σύντομης, της κατεπίγουσας. Ξεκίνησε τον Ιουνιό πέρσι, πρώτη δεκάτου ήταν η προθεσμία για την ε, υποβολή των υποψηφιωτήτων. Ανοιχτήκαν οι φάκελοι, γίνεται τώρα η τελική φάση της αξιολόγησης, οπότε και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση κατά το πρώτο τρίμηνο φέτος. Και θα γίνουν και υπογραφές, τέλος πάντων η ανάθεση της σύμβασης πλαίσιο το επόμενο τρίμηνο. Πέραν τώρα αυτών των ε, δύο βασικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ε, αναγκαίες μεταβολές, τις τροποποίησεις του ισχύοντος συστήματος VIS και το συμμεταυτοποίηση των βιομετρικών στοιχείων που πάει χέρι-χέρι με το VIS. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που θα επιφέρει η εφαρμογή του συστήματος οδοεξόδου, οπότε γι' αυτό και οι τροποποιήσεις θα γίνουν με συγκεκριμένη ε, σύμβαση και η εφαρμογή, η υλοποίηση, από ό,τι προβλέπετε, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, πρώτες μέρες του Απριλίου του 19 ή τέλο πάντων κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Θα πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε την υποδομή επικοινωνίας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα όσα απαιτεί το συστημα εισόδου Αυτά όσον αφορά τις διαδικασίες. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος προηγουμένως. Έχουμε συμβάλει στην υπόθεση των εφαρμοστικών πράξεων. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, όπως αναφέραμε προηγουμένως και όπως προβλέπει το άρθρο 37 παραγραφός 2 τα όργανα διακυβέρνησης που προβλέπονται κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ήδη έχουν συγκροτηθεί. Οπότε έχουμε το Program Management Board που αποτελείται από 10 μέλη το οποίο συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο κανονισμός. Ε, αυτό το συμβούλιο, αυτό το όργανο ας πούμε, εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει το σωστό management κατά την ε, φάση σχεδιασμού και ανάπτυξη του συστήματος και θα υπάρχει συντονισμός ε, μεταξύ κέντρου και κράτων μελών. Ήδη τον Μάιο ε, συνεδρίασε αυτό το όργανο και από τότε μηνιαία συνεδριάζει. παράλληλα με την ε, ομάδα των συμβούλων που συγκροτήθηκε και συνεδρίασε στην Εστονία, στο Ταλίν, στις 5 Ιουνίου, εκεί που είναι η έδρα μας. Εκεί έγιναν οι διορισμοί και από τότε έχουμε έξι συνεδριάσεις κάνει και η επόμενη θα είναι στο Στρασβούργο. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε να δούμε τους εθνικούς ε, εκπροσώπους για όλα τα θέματα θα τα συζητήσουμε και κατόπιν θα αναφέρουμε σχετικώ στα διοικητικά μας όργανα, τα governance bodies. Για όλους όσοι μπλέκονται στο σύστημα παραλίλω, σας ενημερώνω για το εξή. Υπάρχει στενή συνεργασία της υπηρεσία με την ΣΥΠΟΛ και με την Frontex. Οπότε γίνονται τα προπαρασκευαστικά σε σχέση με κάποιες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης που χρειάζονται οι χρήστες του συστήματος ε, εισόδου-εξόδου, ώστε να είναι σε ετοιμότητα για την έναρξη λειτουργίας του. Όλα αυτά ήδη ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο πέρσι. Έχουμε κάνει αξιολόγηση των αναγκών και όλα αυτά πρόκειται οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες να τα επεξεργαστούν και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τέλος αυτού του του ημίνου. Όπως σας προείπα έχουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το σύστημα. Αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από το Management Board, όπως είναι ο κύριος και έχει ήδη αρχίσει αυτή η διαδικασία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτές τις προδιαγραφές επίσημα. Ήδη πέρσι είχαμε μια θετική γνωμοδότηση επίσημη αυτό είναι καλό σημάδι και αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν θα σημειωθούν καθυστερήσει στον προγραμματισμό. Παράλληλα, αυτή η επίσημη διαδικασία ακολουθείται και από το Management Board το δικό μας που έχει δώσει την εντολή να γίνει αυτή η διαδικασία. Και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των αξιολογήσεων στο τέλος του πρώτου τριμήνου φέτος. Τώρα όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, κάποιες λεπτομέρειες, δεν έγιναν τίποτα πληρωμές όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος κατά αυτή την πρώτη περίοδο ενημέρωσης με τις εκθέσεις. Ήδη έχουμε δεσμεύσει πάντως κάποια κονδύλια σχετικά με τον προϋπολογισμό μας και θα λάβετε έναν σχετικό πίνακα στην έκθεση που θα σας ε, διαβιβάσουμε. Αυτά ήθελα να σας ενημερώσω για το σημεσόδεξο. Τώρα για το αίτιας, σε ένα πέντε λεπτά και λιγότερο για να ενημερωθείτε. Υπάρχει το πρόγραμμα και έχουμε τρεις δέσμες, τεχνικές προδιαγραφές, νομικά θέματα, τεχνικά θέματα και συνεχώς προχωρούμε την προπαρασκευή και όπως προηγουμένως γίνονται σε αυτά σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη όσον αφορά την προετοιμασία των εφαρμοστικών πράξεων και συνεχώς γίνεται η διαδικασία των προσλήψεων για περίπου 40 πρόσωπα. Ελπίζουμε φέτος θα ολοκληρωθεί αυτό στο δεύτερο, τρίτο τρίμηνο και επίσης ε, θα γίνει ο διαγωνισμός τέλος του 19 ή αρχάς του 20. Υπάρχει το όργανο διακυβέρνησης και το Management Board θα, θα συνεδριάσει πρώτη φορά 1η Φεβρουαρίου. Και το πρώτο advisory group και για τα δύο συστήματα αιτία και ισοδοξό θα γίνει 14 Τρίτου στο Ταλίν. Οπότε εκεί θα συζητηθούν διάφορα. Προγραμματισμό, συνεργασία με Frontex και Europol, κρατημέλη, όσου εμπλέκονται τέλο πάντων, μηδενικό προπολογισμό ακόμη. Ε, δεν χρειαζόταν να γίνουν τίποτε δαπάνες προς το παρόν. Είμαστε ακόμα στην αρχή και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σύρκο. Ακούγοντάς σας και τους δύο, έχοντας μάλλον ακούσει και τους δύο, ε, είχαμε το χρόνο να σκεφτούμε το τι έχουμε νομοθετήσει σε σχέση με αυτά τα δύο θέματα, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους είναι αυτό που σχετίζεται με την τεχνολογία της πληροφορίας. Και κάνοντας κανείς ένα απολογισμό των έχουν συμβεί σε σχέση με από τη στιγμή που εγκρίναμε αυτά τα δύο συστήματα μέχρι τώρα, βλέπουμε πόσο τεράστιο είναι το σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας παλιότερα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκπρόσωπο του Σιγιου τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για αυτές τι παρουσιάσεις. Ας ακούσουμε και τα μέλη της Επιτροπής μας που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα, τα δύο θέματα. Καταρχήν με την κυρία Γκάλ να ξεκινήσουμε που είναι η συγκέντρια για το αιτία. Κυρία Γκάλ, έχετε το λόγο. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Σούλαν και τον κύριο Σύριγο για την παρουσίασή τους και κυρίως για το πόσο έχουν δουλέψει, για το τι έχουν κάνει. Το project αυτό, οι διαδικασίε είναι πολύ περίπλοκες, γεμάτες με προβλήματα και προκλήσεις. Έχω μια-δυο ερωτήσεις σε σχέση με αυτές ακριβώς τις προκλήσεις και τις απευθύνω και στους δύο σας. Κύριε Σουλών, είπατε ότι το ένα από τα σημεία κλειδιά στην εφαρμογή θα είναι η συνεργασία με, τα, με τις αρχές. Ε, πιστεύετε ότι οι αρχές των κρατών μελών είναι προετοιμασμένες και σε ποιο βαθμό. Προφανώς οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει, αλλά πόσο έχουν προχωρήσει έτσι ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ξέρω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κατεξιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Πιστεύετε όμως ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα μας δυσκολέψουν στο μέλλον και θα καθυστερήσουν τη διαδικασία εφαρμογής του αιτίας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας τρίτες χώρες. Τι αντιδράσεις έχουν σε σχέση με αυτά τα συστήματα. Σε σχέση με αυτά τα δύο συστήματα αιτίας και σύστημα εισόδου-εξόδου. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο, κάποια περίπτωση εξαιτίας αντιδράσεων τρίτων χωρών να πέσουμε έξω στο χρονοδιάγραμμά μας ή στον προγραμματισμό μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Αγκάλ. Σιλβί Θα είμαι πιο σύντομη εγώ. Η κυρία Γκάλ έθεσε το πιο κέριο θέμα που ήθελα και εγώ να θίξω. Θέλω βέβαια να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, δύο συναδέλφους παρεμβαίνοντες. Ε, με τις παρουσιάσεις τους μας κατέδειξαν την περιπλοκότητα του θέματος. Εγώ μιλώ πιο πολύ για το αιτίας γιατί το γνωρίζω καλύτερα. Ε, και εγώ έχω την ίδια ερώτηση με, την, με αυτήν της Κίνγκα Γκάλ. θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Πόσο έχουν προχωρήσει οι προετοιμασίες στα κράτη-μέλη στο ζήτημα του αιτίας, γιατί θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια για το Μητρό Επιβατών μας είχε ζητηθεί να βιαστούμε πάρα πολύ, αλλά καθυστέρησε τελικά εξαιτία προβλημάτων στην τελική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Οπότε ήθελα να, να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα από πλευρά των κρατών μελών. Προέδρο Μπάρμπαρα Κουτζίσκα. Ε, δύο ερωτήσει για τον κύριο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, στον κανονισμό η Γιουλίζα είχε προβλεφθεί μια διάταξη για την ε, προστασία προσθήκη, για τη διεύρυνση ε, της έδρας σας στο Στρασβούργο, επειδή αυτή τη στιγμή η έδρα σας δεν έχει επαρκή υποδομή. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το θέμα. Μετά στην έκθεσή σας για την ανάπτυξη του συστήματος εισόδου-εξόδου αναφέρεται ότι ε, πρόσθετες αλλαγές, ίσως χρειαστούν πρόσθετες, ίσως τα κράτη-μέλη ζητήσουν μάλλον πρόσθετες αλλαγές στην, ε, στο κανονιστικό πλαίσιο. Ε, πώς θα καταφέρουμε τέτοιες αλλαγές να μην καθυστερήσουν το χρονοδιάγραμμα. Τέλος, για το αιτίας. Πού βρίσκεται η εφαρμογή του. Έχουν προκύψει κάποια απρόβλεπτα εμπόδια ή όλα πηγαίνουν ομαλά, βαίνουν ομαλώς. Ευχαριστώ. Ο κ. Φρανς. Γεια σα. Καλή σα μέρα. Μία ερώτηση για το Ιουλίζα. Το Ιουλίζα ε, συνεργάζεται και με εταιρείε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που συλλέγουν δεδομένα. πώ βεβαιώνεστε, πώ εγγυάστε την εμπιστευτικότητα αυτών των στοιχείων και ότι δεν θα φτάσουν σε χέρια που δεν, τα, δεν θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ελαιοπρόεδρος Καλός Κουέλιο. Ο κ. Δίαθ Μέρα δεν κατάφερε να φτάσει στις Βρυξέλλες, οπότε μου ζήτησε να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές. Θέλει να υπογραμμίσει την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στην Ιουλίζα, την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην σημασία της διαφάνειας για το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τη διαδικασία εφαρμογή των, των πληροφορικών συστημάτων. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, καλωσορίζουμε την δημιουργία των διαφόρων ομάδων και οργάνων που θα εξασφαλίσουν μια σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή σύμφωνα με τα καθήκοντά του. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό, σήμερα μιλούμε για το έργο που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά μην ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα κράτη-μέλη. Υπ' αυτή την έννοια, ο κ. Διαντεμέρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Η Κομισιόν σκοπεύει να λάβει κάποια πρωτοβουλία για να παρακολουθήσει τι προετοιμασίε που γίνονται στα κράτη-μέλη, προκειμένου να εγγυηθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα είναι έτοιμα τη στιγμή που η Ιουλίζα θα έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου αν καθυστερούν κάποια κράτη-μέλη να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε. Ένα από τα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι επίση η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προπολισμού. Η Γιουρίζα μα ενημέρωσε για τις διάφορες διαδικασίες προσλήψεων και καλωσορίζουμε τη διαφάνεια αυτή. Στις 7 ε, Ιανουαρίου η Κομισιόν υπέβαλε μια νέα νομοθετική πράξη που τροποποιεί τον αιτία προκειμένου να συνδεθεί με τα άλλα συστήματα, για παράδειγμα το σύστημα εισόδων-εξόδων. Ο κ. Διαδεμέρα θεωρεί ότι για την Ιουλίζα είναι πολύ σημαντικό να έχει τον κατάλληλο προπολογισμό προκειμένου αυτή η καινούργια πρόταση της Κομισιόν να μην επιδράσει αρνητικά στη σωστή εφαρμογή του των συστημάτων αυτών. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σαφής οι ε, ερωτήσεις σας, οπότε θα επιστρέψουμε στους συναδέλφους της Κομισιόν και της Ιουλίζα. Με συντομία όμως παρακαλώ. Καταρχήν ο κύριος Σουλών. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Πράγματι, η Κομισιόν ξεκίνησε ήδη να παρακολουθεί τις ε, προετοιμασίες των κρατών μελών. Ξεκινήσαμε ένα γύρο πρωτεύουσών και θα τον συνεχίσουμε κατά τη διάρκεια του τρέχοντο έτους. Ήδη έχουμε επισκεφθεί 12 πρωτεύουσε και έχουμε συναντήσει τις ε, αρμόδιες αρχές παρακολουθώντας και το, τις εξελίξεις του κανονισμούς που συζητώνται αυτή τη στιγμή με τους συνσηγητές. Στα αυτές μας επισκέψεις καταρχήν ενημερώσαμε τα κράτη-μέλη, ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη για τις δικές μας Προσδοκίε ό,τι αφορά την ετοιμασία του. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να μετρήσουμε το στάδιο, να ε, εντοπίσουμε το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι προετοιμασίε. Συγκρίνοντας το τι έχει γίνει στα κράτη-μέλη, συλλέγοντα τι βέλτιστε πρακτικέ, ε, ενημερώνοντα τα κράτη-μέλη για τι βέλτιστε πρακτικέ, διότι ε, χρειάζεται όλοι να είναι στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε μάλιστα και ένα βαθμολόγιο έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε το στάδιο προετοιμασίας του ενός και του άλλου. Το σημαντικό είναι όμως όλα τα κρατη να είναι έτοιμα την κατάλληλη στιγμή. Εν τω μεταξύ και στους δύο κανονισμούς υπάρχουν διατάξεις που λένε ότι το σύστημα, τα συστήματα δεν θα αρχίσουν να λειτουργούν αν δεν έχουν δηλώσει όλα τα κράτη-μέλη τη λήξη των προετοιμασία της προετοιμασίας τους, όπως ακριβώς λέει ο κανονισμός. Το σε αφορά τις αντιδράσεις των τρίτων χωρών. Έχουμε πιο πολλά αιτήματα πληροφόρησης και λιγότερες αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή τα, οι τρίτες χώρες προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα λειτουργήσει το σύστημα για τους ε, ταξιδιώτες. Ιδιαίτερα ε, οι διευκρινήσει ζητούνται από tour operators ή από ταξιδιωτικά γραφεία. Οπότε έχουμε ετοιμάσει πακέτα πληροφοριών, kit, τα οποία μοιράζουμε μέσω των διπλωματικών μας ε, αποστολών στις τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του αιτία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέω ο κύριε Σίγου, για την Ιουλίζα. Σε ό,τι το θέμα της ικανότητας του κέντρου δεδομένων μας, του data center. Ξέρουμε ότι το σύστημα εισόδου-εξόδου έχει πολύ υψηλέ απαιτήσει σε ό,τι αφορά την απόδοση και τη διαθεσιμότητά του. Οπότε ήδη αναζητούμε αρχιτεκτονικές λύσεις ε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο που αυτές οι καινούργιε απαιτήσει θα έχουν σε εμά. Είμαστε σε επαφή με την Κομισιόν για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Εξετάζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα γίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα του αιτίας και του κατά πόσον η εφαρμογή γίνεται με ομαλό τρόπο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε στενή επαφή με τη Frontex, τη Europol, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, όλους του ενδιαφερόμενους και σε συνεργασία με αυτού εντοπίζουμε ε, τα στοιχεία που χρειάζεται να έχουν οι κατοξιοδότης πράξεις και οι εκταλιστικές πράξεις. Έχουμε τρεις ε, παράλληλες ε, διαδικασίες, ε, προσλήψεις, τεχνικές προδιαφές. Σας είπα, σας τα είπα αυτά. Όλα αυτά πηγαίνουν καλά, βαίνουν ομαλώς. Τώρα σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που μπορεί να ζητήσουν τα κράτη-μέλη. Να, να επαναλάβω ότι έχουμε ξεκινήσει από το 2016 συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και μάλιστα λεπτομερείς συζητήσεις για διάφορα τεχνικά θέματα και τα έχουμε συμφωνήσει. Όλα αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί και θα συμπεριληφθούν και στις ε, εφαρμοστικές πράξεις οι οποίες θα εκδοθούν στο μέλλον. Και στις ε, δημοπρατήσεις που κάνουμε προβλέπουμε τεχνικές προδιαγραφές που έχουν σχέση με την ε, μηχανή workflow, όπως είπα και προηγουμένως. Οπότε οι προσκλήσεις διαγωνισμού διαγωνισμούς και οι τεχνικές προδιαφές που έχουμε περιγράφουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ζήτησαν τα κράτη-μέλη. Αν αργότερα ζητήσουν κάτι παραπάνω, διαθέτουμε διαδικασίες διαχείρισης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα αιτήματα και να ικανοποιηθούν. Όμως μετά την λεπτομερή διαδικασία που έχει λάβει χώρα ήδη δεν προβλέπω να υπάρχουν τέτοιου αιτήματα από πλευρά των κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των δεδομένων σε ξένε εταιρείε. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω το εξή. Οι εταιρείε δεν έχουν πρόσβαση σε κανενός είδου δεδομένο. Δεύτερον, δεν υπογράφουμε συμβάσει με ξένες εταιρείε. Αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλάμε για μια νομοθεσία που εφαρμόζεται σε εταιρείε συνολικά και στην Ευρώπη ιδιαίτερως. Αυτό τι την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εφαρμόζουμε. Ε, νομίζω ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν ξέχασα κάποια παρακαλώ πολύ πέστε μου το. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ιουλίζα και την Κομισιόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους που παρακολουθούν στενά αυτό το πολύ σημαντικό project. Το θέμα αυτό θα παρακολουθεί και από το καινούριο κοινοβούλιο προφανώς. Εμείς εδώ μεταξύ κάνουμε τη δουλειά μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ε, σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Eurojust και Γεωργίας έχει μια σειρά συμφωνίων με τρίτε χώρε η Eurojust. Πρόσφατα υπογράφηκε μια συμφωνία με την Αλβανία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία διαβούλευση. Το Κοινοβούλιο έχει μια προθεσμία τριών μηνών για να εκφέρει γνωμοδότηση. Η προθεσμία λύγει στι 16 Φεβρουαρίου και μπορούμε μόνο ή να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε το περιεχόμενο τη συμφωνία. Εξαιτία του επίγοντο τη διαδικασία, οι συντονιστέ αποφάσισαν μια απλοπλουστευμένη διαδικασία, δηλαδή να μην υποβληθεί καμία τροπολογία. Ε, μόνο έτσι κι αλλιώ μόνο ε, διαδικαστικές τροπολογίες ήταν ε, δυνατόν να καταληθούν. Θέλω να δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στον εισηγητή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Κλοντ, θα είμαι συντομοτάτη σχετικά με την ε, συμφωνία σκοπός της οποίας είναι η συνεργασία κατά την καταπολέμηση βαριάς εγκληματικότητας και ιδίως της οργανωμένης και της τρομοκρατίας. Επιτρέπει την ανταλλαγή αξιωματούχων συνδέσμων, ανταλλαγή πληροφοριών και δημιουργία σημείων επαφής. Η Συμφωνία Συνεργασίας Eurojust Γεωργίας ακολουθεί το πρότυπο άλλων συμφωνιών που διαθέτουμε. Η Eurojust ήδη έχει με την Μακεδονία, τις Ηνωμένε Πολιτείες, Νορβηγία, Ελβετία και πρόσφατα, όπως είπες και εσύ, Κλοντ, με την Αλβανία. Τέτοιες, έχει συνάψει λοιπόν τέτοιες συμφωνίες. Θεωρώ ότι είναι καλή η συμφωνία και σημαντική, διότι Υπάρχουν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στις χώρες μέλη και προέρχονται από την χώρα αυτή. Γνωρίζουμε ότι η Γεωργία είναι επίσης μια χώρα η οποία βγαίνει από μια σύγκρουση, έχει διαθέσιμο μεγάλο αριθμό όπλων που κυκλοφορούν και ενδεχομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε λαθρεμπόριο όπλων. Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, κατάργηση των προξενικών θεωρήσεων δηλώνει ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος από την Γεωργία εξακολουθούν να είναι από τις πιο συχνά και πυκνά συναντώμενες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή τους σε βαριά εγκλήματα. Εν ώψη αυτού του ιστορικού η συμφωνία μεταξύ Eurojust και Γεωργίας αναμένεται να διευκολύνει την συνεργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο και είναι προ το συμφέρον και τη Γεωργία και των χωρών μελών τη Ένωση, διότι η οργανωμένη, το οργανωμένο μάλλον έγκλημα είναι πολύ καλά δικτυωμένο. Το 2017 συνήψε σχετική συμφωνία η Ευρωπόλ. Έτσι λοιπόν η συμφωνία τώρα της Eurojust είναι στην πραγματικότητα μια πολύ σκόπιμη συμπλήρωση. Για θέματα τώρα προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία για την ίδρυση της Eurojust, τέτοιου είδους συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Eurojust και τρίτων χωρών, που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα, μπορούν να συνάπτονται μόνο όταν υπάρχει εγγυημένο ένα επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εδώ η κοινή αρχή η αρμόδια αρχή της Eurojust δηλαδή, διαπιστώνει, έχει μάλλον εκδώσει θετική γνωμοδότηση και έχει δηλώσει ταυτόχρονα ότι σχετικά με το άρθρο 17 του σχεδίου της ε, συμφωνίας δεν έχει λάβει καμιά κοινοποίηση, μάλλον δεν προβλέπεται κοινοποίηση για θέματα προσβολής προσωπικών δεδομένων μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή Eurojust και Γεωργία. Γι' αυτό και προτείνεται το στοιχείο αυτό να συζητείτε στη διάρκεια των τακτικών συνεδριάσεων με Γεωργιανού ομολόγους τους, να συζητείτε δηλαδή μεταξύ Ευρωπαίων και Γεωργιανών αρμοδιών. Εν το συνόλο, όπως είπες και εσύ αγαπητέ πρόεδρε, Ούτω ή άλλω εμεί μπορούμε μόνο να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο τη συμφωνία. Όμω, από την άποψή μου, θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν καλώ και θα πρέπει να εγκρίνουμε και μάλιστα ε, σύντομα, διότι όπω ε, τόνισε και εσύ, ο χρόνο πιέζει. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς δεν είναι εδώ από τους σκιώδες. Αλλά αν δεν μπορεί να το κάποιο κύριε Φράντ, έχετε το λόγο. Συμφωνούμε, συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε με, την, ε, με το σχέδιο. Α, συντομότατο. Παρά ήταν σύντομο. Όχι, δεν θα σα πιέζω σε σχέση με το πόσο θα μιλήσετε, πόσο θα αγορεύσετε, θα είναι κακό και αντιδημοκρατικό. Οπότε τώρα Φαντάζομαι. 29 δεύτερο θα δώσουν το πράσινο φω. Πάλι δεν έπρεπε να το προκαταλαμβάνω. Ωραία, ωραία, ολοκληρώσαμε με το θέμα και στι 29 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε και θα πάει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου το θέμα. Και τώρα πάμε στο 26. Θέσπιση Ταμείου Ιστορική Ασφάλεια. Εξέταση και κειμένου. Ε, η συγγήτρια είναι η Μονικά Χόλμαρ, την έχουμε εδώ και πάλι συμπαθώτε με μια που έχουμε αργήσει. Όλα τα θέματα έχουν πάει πίσω, εγώ φταίω. Όπω έλεγα, είναι συζήτηση του σχεδίου κειμένου για αυτή την νομοθετική πρόταση που αφορά το Ταμείο Ιστορική Ασφάλεια. Οπότε σου με το λόγο τώρα για να μα τα εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κλοντ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω και εγώ να συντομεύσω κάπως, διότι για το ESF συνεργάστηκαν όλοι οι συναρμόδιοι εισηγητές και σκιώδεις πάρα πολύ καλά. Ιδίω εγκύψαμε σε ορισμένε τροπολογίε, για τι οποίε άλλωστε ευχαριστώ του συναδέλφου, διότι είναι και ακριβώ διατυπωμένε και καινοτόμε και αντιμετωπίζουν σωστά ε, το θέμα. Για παράδειγμα την προώθηση συνεργασίας με υπηρεσίες πληροφοριών για τη δημιουργία ε, μιας ευρωπαϊκής ε, υπηρεσίας πληροφοριών, τροπολογία των φιλελευθέρων. Το κρίσιμο ερώτημα τι σημαίνει η συμπερίληψη του ιδιωτικού τομέα, διότι δεν θελήσαμε ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει καθήκοντα του δημοσίου, Όμω προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε τα πράγματα εδώ. Η κυρία Σεσίλ Κιένγκε ε, ε μας ε, συνεργάστηκε και μα διευκόλυνε για αυτή την διευκρίνηση, διότι σημαντικά καθήκοντα τη της δημοσίας αρχής δεν θέλαμε να αναλυθούν από ε, ιδιωτικές δομές. Θέλουμε να περιοριστούν να περιοριστεί η συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα μόνο όπου αυτή είναι απαραίτητη. Τρίτο, για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και τους ε, συναρμοδίους ε, ε, διεθνείς οργανισμούς, συμφωνήσαμε εν τέλει ότι στοχεύουμε ιδίως στην εργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ότι η σχετική συνεργασία θα γίνεται μόνο υπό τους όρους του ESF, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφαλείας του Ταμείου Εσωτερικής ασφάλεια Πιο σωστά. Και για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρε θα περιοριστούμε στα πλέον σημαντικά θέματα. Τέλος, προσπαθήσαμε να καταστήσουμε επίσης σαφές ένα άλλο θέμα. Εντός των πλαισίων των δομών ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχουν διαφορετικές δομές και ορισμένε χώρε μέλη στον τομέα ασφαλείας διαθέτουν δομές και οργανώσεις που συμπεριλαμβάνουν και τον στρατιωτικό ή υπόκεινται στον στρατιωτικό τομέα ή στο Υπουργείο Αμήνης και επιτρέπουν και συμμετοχή στρατιωτικών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, όπως για παράδειγμα καταπολέμηση τρομοκρατίας, όπως ε, βλέπουμε και εδώ στο Βέλγιο. Που δεν είναι το συνηθές, αλλά συμβαίνει. Στην Ιταλία και στην Ισπανία έχετε παρόμοιες δομές όπως η Guardia Civil, η ε, Ισπανική Πολιτοφυλακή, που είναι ε, πλέον ένα ε, ιστορικό δεδομένο. Αποφασίσαμε ότι με το Ταμείο αυτό δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε δράσεις εκτός Ευρώπης, για παράδειγμα, ειρηνευτικές δραστηριότητες στο Μάλι. Είπαμε ότι θα παραμείνουμε εντός συνόρων. Και έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω εν τέλει τις και τους σκιώδης για την επικοδομητική συνεργασία. Προσπαθούμε και για τα διάφορα οριζόντια θέματα τα οποία υπερβαίνουν ας πούμε και τα όρια του Ταμείου να συνεννοηθούμε και ε, με αυτούς που διαχειρίζονται τα άλλα ταμεία, όπως για παράδειγμα άσυλο μετανάστευση ή ε, για θέματα προξενικών θεωρήσεων, ώστε να μην καταλήξουμε σε δομέ οι οποίες ενδέχεται να δείχνουν και αντιφάσει μεταξύ τους. Με την έννοια αυτή λοιπόν ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ ε, όλος ιδιαίτερα στην Γραμματεία για την στήριξη που έδωσε στην εργασία μας και ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε, να υπερψηφίσουμε μάλλον με μεγάλη πλειοψηφία τον, ε, ε τον, την δομή αυτή του Ταμείου Συντηρικής Ασφαλείας. Ευχαριστώ. Σεσίλ Κιένγκε, επιθυμείτε να λάβετε το λόγο, όσοι Σκιώδης. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ να ευχαριστήσω την Μολίκα Χολμάγερ, την εισηγήτρια. Γιατί έδειξε μεγάλη πρόθεση συμβιβασμού, πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα. Πάρα πολύ έχουμε προσπαθήσει για να αναζητήσουμε την επίτευξη συμβιβασμού και τελικά να περάσει το σχέδιο κανονισμού μέχρι το τέλος αυτής της θητείας. Με, μια πρώτη ματιά των προτάσεων συμβασμού μπορέσαμε να αναλύσουμε και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο το κείμενο και εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι θετικά όσον αφορά αυτές τις πρώτες προτάσεις που έχω λάβει και με την ε, εισηγήτρια αλλά και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Είπαμε ότι θα πρέπει ε, να προσθέσουμε και την βία, η τρομοκρατία, την ριζοσπαστικοποίηση, ε, την έλλειψη ανεκτικότητος στους στόχους. Και επίσης όσον αφορά την κατανομή του κόστους έχουμε κάνει προτάσεις στις τροπολογίες μας. Είμαι βέβαιη ότι όλα αυτά που κάναμε θα οδηγήσουν στο να μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας την διαδικασία και είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μας πολιτική ομάδα. Θα δούμε θα γίνει και με τη συμμετοχή των τρίτων ε, χωρών. Άκουσε τη γνώμη της εισηγήτριας, της, ε, το ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών και των ε, στρατιωτικών υπηρεσιών για να έχουμε έτσι τελικά αυτό το ταμείο να εξυπηρετήσει τους σκοπούς που πέπρονται. Οπότε ελπίζω όπως έλεγα θα καταλήξουμε σε συμβασμό με την εισηγητρία όλους. Τους ευχαριστώ και την εισηγήτρια και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε σας, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Φραντς, από τους άλλους σκιώδες. Κυρία Χολμάιερ, σας ευχαριστώ και εγώ για την ε, πολύ θετική επικοδομητική συνεργασία και εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι υποστηρίξατε πολλές από τις τροπολογίες μας και ιδίως όσον αφορά την περαιτέρω κατάρτιση και ευαισθητοποίηση για θέματα ε, ρατσισμού των αστυνομικών δυνάμεων και το πρόγραμμα που προτείναμε ανταλλαγή νεαρών αστυνομικών υπαλλήλων, όπως γίνεται ας πούμε με το έρασμο για του σπουδαστέ, θα συμβάλλει ότι θα βελτιωθεί η διαμεθοριακή συνεργασία. Χρειάζεται ακόμη δουλειά βέβαια για τις συμβαστικές τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πλήρες πράσινο φως. Για τον ορισμό της κυβερνοεγκληματικότητας υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά ακόμη θεωρούμε ότι ακόμα ο ορισμός του κυβερνοεγκλήματος δεν είναι αρκετά σαφής. Διότι μεταβάλλεται κιόλα. Με κριτικό πνεύμα εξετάζουμε επίσης τις δραστηριότητες όπου συμμετέχει και ο στρατός. Θα πρέπει στο κείμενο να είναι σαφέστερη διατύπωση ότι πρόκειται μόνο για αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων. Το ίδιο η συμπερίληψη των μυστικών υπηρεσιών στην χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ιστορικής ασφαλεία. Εμεί θέλουμε να το αποκλείσουμε αυτό. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των χωρών μελών και ο δαμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει επίση να υπαγορεύεται στι χώρε μέλη ότι θα πρέπει να διατηρούν ένα αποθεματικό στον προπολογισμό του Ταμείου Ιστορική Ασφαλεία για τη χρηματοδότηση μυστικών υπηρεσιών και εμείς, η ομάδα των Πρασίνων δηλαδή, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε εφόσον γίνουν ακόμη κάποια βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φραντς. Άλλος κανείς? Νόμιζα πως κάτι θέλατε να πείτε ε, ίσως ε, ήμουν υπερβολικός όμως. Κύριε Σιγητά, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι τους και Σιγητές. Κάναμε πολύ και σκληρή δουλειά. Θα επανεξετάσουμε τη διατύπωση για το στρατιωτικό τομέα. Η νομική υπηρεσία μας λέει ότι ο ορισμός είναι σαφής. Θα το ξαναδούμε όμως. Εμείς συμφωνούμε πάντως ότι ο ESF θα επιτρέπει μόνο παρεμβάσεις στο εσωτερικό. Έχουμε και διαφορετικές παραδόσεις στις διάφορες χώρες μέλη. Όπως είπαμε, η Guardia Civil των Ισπανών είναι στρατιωτική δομή, είναι αμυντική δομή και υπάγεται στο ε, Υπουργείο Αμήνης. Είναι έτσι. Δεν πρόκειται όμως για επεμβάσεις στην αλλοδαπή. Αλλά όπω είδαμε, α πούμε, χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των τρομοκρατών στον Μπακτακλάν, στη Γαλλία, στο Βέλγιο για την ε, εγγύηση τη εσωτερική ασφάλεια. Όπω βλέπουμε στην Ιταλία και η Ισπανία με τι ιστορικέ αυτέ ε, στρατιωτικέ δομέ που ε, χρησιμοποιείται για την ε, δημόσια ασφάλεια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και μπορεί η συνδρομή του για την αντιμετώπιση τη τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματο είναι πολύ σημαντική. Όμω, ιστορικά έχουν διαφορετικέ δομέ. Εμεί στη Γερμανία δεν έχουμε τέτοια δομή. Παριμήν τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα και διακριτά. με πολύ διαφορετικές οι δομές. Όμως ο ESF προβλέπει μόνο κατάλογο καθηκόντων, ώστε επεμβάσει στο εξωτερικό, στην αλλοδαπή δηλαδή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είναι δυνατέ ούτω ή άλλω και με κανένα τρόπο δεν θα καλύπτονται χρηματοδοτικά από το, από το Ταμείο Εσωτερική Ασφαλεία. Θα το καταστήσουμε ακόμα σαφέστερο όμω ώστε κανείς να μην μπορεί να παρανοήσει και να μπορέσουν όλοι τελικώς να συμφωνήσουν. Ότι δεν θέλουμε δηλαδή να αναμειγνύεται το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας με κανένα τρόπο σε εξωτερικές, εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Επικράτειας θέματα. Σε αυτό είμαστε απολύτω σύμφωνοι όλες οι πολιτικές ομάδες. Το δεύτερο για το Cyber Enabled Crime για το Cyber Enabled Crime, λοιπόν, τονίζω ότι πρόκειται ιδίω για είδη εγκληματικότητα και αυτό ε, πλήττει όλε τι χώρε μέλη και έχουν του ίδιου ορισμού. Ο ορισμό είναι σκόπιμο. Ε, ανταποκρίνεται στο στόχο του, δηλαδή όπω είναι. Θα πρέπει να δούμε, αν, ας πούμε, πάρουμε μια περίπτωση απάτης. Μια περίπτωση απάτης εάν φύγει ένα πρόσωπο κάπου, έχει διαφορετική άξια από το εάν γίνεται μέσω του διαδικτύου cyber-enabled δηλαδή, που έχει μετά δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της απάτης αυτής ε, παντού. Το ίδιο η ε, γενετήσια κατάχρηση παιδιών, που είναι επίσης ε, μια βαρβαρότητα η οποία διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου και η οποία βέβαια διαδίδεται με βάρβαρο τρόπο και ε, διαφεύγει της ε, ε, δύσκολο να διωχθούν όλοι τελικώς οι, ανα, οι αναμειγνιόμενοι. Και μέσω του διαδικτύου είδαμε ε, σημαντική ενίσχυση της εγκληματικότητας σε διάφορους τομείς που πριν υπήρχαν τα εγκλήματα αυτά αλλά σε μικρότερη έκταση. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι Αυτό, αυτή η διάκριση και αυτοί οι ορισμοί μας φαίνονται πάρα πολύ σημαντικοί για να αποφεύγεται οποιαδήποτε ε, σύγχυση. Τέλος, για τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είχαμε συμφωνήσει και η νομική υπηρεσία έτσι μας το εξήγησε και το όρισε ότι πρόκειται μοναχά για συνεργασία. Δεν τίθεται θέμα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκούμε επιρροή στις δομές των υπηρεσιών ασφαλείας. Ούτε είναι και καθήκον του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας να χρηματοδοτεί υπηρεσίες πληροφοριών. Όχι. Πρόκειται μόνο για ανταλλαγή πληροφοριών και για το είδος της ανταλλαγής πληροφοριών. Πρόκειται για την βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Βαρέως οργανωμένου εγκλήματος. Ο ορισμό τον οποίο πρότεινε ο Λουί Μισελ είναι αρκετά ακριβή. Σας παρακαλώ εξετάστε και πάλι τις τροπολογίες οι οποίε μάλιστα κατατέθηκαν χθε, ορισμένε εξ αυτών, διότι θεωρώ ότι η πρόταση του Λουί Μισελ την οποία στηρίζουμε και εμεί αλλά και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, είναι σαφώ ορισμένη και δεν παρεμβαίνει σε ενδεχόμενε εσωτερικές δομές. Πρόκειται λοιπόν αυστηρά για ευρωπαϊκή ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς καμία ανάμειξη στην εσωτερική ασφάλεια. Σε εσωτερικά θέματα δηλαδή ε, ε, υπηρεσιών ασφαλείας. Το καλύτερο είναι νομίζω να το ξαναδούμε διμερώς, να ε, δούμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, για παράδειγμα παιδική πορνογραφία, να καθίσουμε να τα δούμε πάλι αυτά και να ξεδιαλύνουμε ορισμένα τεχνικά ερωτήματα όπου νομίζω μπορούμε να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις και νομίζω βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή. Αν υπάρχει ακόμα ανάγκη συζητήσεως δηλαδή ή ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ Μόνικα. Και εσύ έχεις κάνει πολύ δουλειά σε αυτό το θέμα και οι σκιώδεις ακούγανε με προσοχή όλα όσα έλεγες. Ωραία, θα ξανασυζητηθεί το θέμα. Η, η ψηφοφορία στην Λίμπη θα λάβει χώρα 18-19 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και εσένα και τους σκιώδης ηγητές. Πράγμα στο σημείο 24 και 25 μαζί, κοινή συζήτηση. Παρουσίαση από πλευρά Επιτροπής, δύο καινούργια ανακοινώσεων στο θέμα της κοινή πολιτικής θεωρήσεων. Πρώτο, ε, κατάσταση μη αμοιβαιότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ΟΠΑ και τη Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, πέντε κράτη-μέλη, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η αμοιβαιότητα. Δεύτερο έγγραφο, έκθεση για το μηχανισμό αναστολή απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση. για το πρώτο θέμα, όπω γνωρίζετε, για την μία αμοιβαιότητα δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στην Επιτροπή μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εκφέρει την άποψή του για την υποχρέωση τη Κομισιόν να υιοθετήσει μία κατεξοδότηση πράξη, οπότε υπογρα... Υπογρα... Ε, λαμβάνουμε γνώση των προσπαθειών της Κομισιόν για να επιληθεί το θέμα. Ε, επιμένουμε στεναρά να επιτευχθεί η αμοιβαιότητα, την οποία είχε ε, πει η Κομισιόν αλλά και η Αυστριακή Προεδρία ότι θα εξασφαλιστεί. Έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον στις 9 Νοεμβρίου 2018 μια υπουργική συνάντηση. Ε, μετά από αυτήν τα τα, η κοινή ανακοίνωση ε, που εκδόθηκε, ε, μας κοινοποιήθηκε και την έχετε, τα πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ανέφερα, τα μεταχείριζε οι Ηνωμένες Πολιτείες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, διότι δεν τα εξαιρεί από ε, δεν εξαιρεί τους πολίτες τους από την ε, διευκόλυνση που έχει δώσει σε σχέση με τις θεωρήσεις στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των υποχρεώσεων της Κομισιόν, που είναι θεσμικό θέμα και καλώς ορίζω την Κομισιόν, ε, ε πολύ καλό το timing, φτάσατε στην ώρα σας. Η άποψη επιτροπή είναι ότι η Κομισιόν έχει υποχρέωση να υιοθετήσει κατεξοδότηση πράξη να ε, ε, μια ε, κατεξοδότηση πράξη προκειμένου να αναστείλει την απαλλαγή από την έκθεση θεωρήσεων για τους Αμερικανούς υπηκός που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Στο θέμα των θεωρήσεων γίνονται πολλές συζητήσεις και τριμερείς διάλογοι. Θα πρέπει να ληφθεί, να ληφθεί υπόψη το θέμα της αμοιότητας σε αυτούς Σαν να την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, σαν να έχουμε ξαναπεί τα ίδια, déjà vu. Καλό είναι όμως να επαναλαμβάνουμε μερικά πράγματα για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό έκανα και εγώ τώρα. Μπορώ να κάνω εγώ την παρουσίαση εκ μέρου σα και κομισιόν, γιατί αν θέλετε. Ε, εντάξει, αστείευομαι. Δεν ξέρω πώ θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να μην επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα. Τέλο πάντων, είμαστε στο τέλος τη μα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η Κομισιόν. Ευχαριστούμε που ήρθατε, έτσι κι αλλιώς. Έχετε το λόγο, κύριε Μίτσελ. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που επιστρέφω. Άκουσα και το θέμα το, της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τη χρηματοδότησή του. Χαίρομαι ε, που θα εκδώσετε ε, εκθεσία 18 και για 19 και μπορώ να πω ότι με τα όσα άκουσα από την συγκήτρια ε, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το θέμα της ε, έλλειψης αμοιβαιότητας. Πρόεδρε, εσείς γνωρίζετε πιο πολλά από μένα. Έχετε εδώ στο Κοινοβούλιο συζητήσει το θέμα και πέρσι. Να σας πω εγώ τι έχει συμβεί τους τελευταίους 3-4 μήνες. Επιπλέον της έκθεσης που περιλάβαμε στο ανακοινωθέν μας στις, ε, το Δεκέμβρη, στις 19 Δεκεμβρίου. Συνεχίστηκαν οι συζητήσεις και συνεχίζονται ακόμα με τις ΗΠΑ για το πώς μπορούμε να πετύχουμε την αμοιβαιότητα, να πετύχουμε δηλαδή τον στόχο μας έτσι ώστε ε, και τα πέντε αυτά κράτη-μέλη να μπορούν να κυκλοφορούν και να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ χωρίς θεωρήσεις. Οι συζητήσει τι οποίε τουλάχιστον εγώ ήμουν παρούσα στι ΗΠΑ με τον Επίτροπο αλλά και μόνη μου με τους ε, συνεργάτες μας εκεί, ε, κατέδειξαν ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία ε, ταξιδιού χωρίς ε, θεώρηση και σε αυτά τα πέντε Και στις συζητήσεις με τον πρέσβη εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και εκεί προσπαθούμε να τους ζητήσουμε, τους ζητάμε βασικά, ε, στοιχεία για, το, για τα ποσοστά ε, απορρίψεων. Μόνο η Κύπρος είναι κάτω από το μεσόρο. Τα άλλα κράτη-μέλη είναι πάνω από το μεσόρο. Εγώ αυτό που ήθελα να μου πούν είναι ποια είναι ακριβώς τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματά τους. Όμως ε, αυτό που λένε οι ίδιοι είναι ότι χρειάζεται να κάνουν μια νομοθετική αλλαγή για τα ποσοστά. Από πλευράς Κομισιών προσπαθούμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να δουλέψουμε, δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας. Και θα ήθελα να σας ζητήσω σε οποιασδήποτε επαφές με τις ΗΠΑ, σε οποιασδήποτε επισκέψεις σας, να πιέζετε κι εσείς όσο πιέζουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω γιατί η Κομισιόν πιστεύει πως δεν πρέπει να δράσουμε με αμοιβαιότητα. Με, δεν πρέπει να την αρχή της αμοιβαιότητας στο συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε διμερός, πολυμερός και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Η έκθεση που υποβάλαμε λέει με άλλα λόγια αυτά ακριβώ που είπα και εγώ τώρα. Την, ε, τον επόμενο μήνα έχουμε ξανά συνάντηση, πάντα βάζουμε το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη, πιέζουμε, οπότε το μόνο που να σας πω είναι ότι εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο έργο μας να πετύχουμε την αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων και για τις πέντε αυτές χώρες και συνεργαζόμαστε και με τα πέντε κράτη-μέλη και με τις ΗΠΑ. Αυτά. Πρόεδρος. Α, μας ενημερώσετε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Πολύ ωραία γιατί είναι το τέλος της θητείας και προχωράμε σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Όμως το θέμα αυτό έχει κολλήσει, κρεμεί. Είναι όμως σε η θέση του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι είναι σοβαρή Τι να σας πω, κάθομαι και σκέφτομαι τι, τι, τι καινούργια προσέγγιση μπορεί να έχουμε. Παραδοσιακά σας πιέζω σχετικά με αυτό. Αλλά οι Αμερικανοί λένε ότι το State Department λέει όχι σε πάρα πολλές αιτήσει χωρίς αυτό να έχει κάποια λογική. Ε, γιατί να μην έχουν ε, την ειλικρία να πούνε ότι θέλουμε κάποιες χώρες να είναι χώρες δεύτερης κατηγορίας. Και όσο και αν αυτό δεν στέκει, ε, από την άλλη είναι γεγονό. Πάρα πολύ καιρό. Και έρχεται το τέλος της θητείας μας. Δεν στέκει, δεν στέκει κάτι τέτοιο. Τα ξέρουμε καλά. Ξέρουμε ακριβώ ποια είναι η θέση του State Department. Και δεν είναι λογικό αυτό που κάνουμε. Γιατί λένε τόσα όχι. Α, και στην Κύπρο ακόμα. δεικτικά το λέω. Γι' αυτό σας λέω. Όλοι τους αυτή η στάση είναι λογική. Οπότε και εμείς τι να κάνουμε. Και γι' αυτό και επανερχόμαστε στο θέμα της δικής σας ευθύνης. Τώρα, τώρα να δείτε τι θα ακούσετε από τους βουλευτές. Τα έχω πει στον αρμόδιο επίτροπο επανειλημμένα. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να προχωρήσω. Και όλα αυτά σας τα λέω πριν εξαπολύσω εναντίον σας τους βουλευτές. Όχι. Ε, ποτέ δεν ήμουν απότομος προς εσάς, αντίθετα από τους Αμερικανούς, ναι. Γιατί όλες αυτές οι αρνήσεις είναι προσβλητικές. Ε, ας ήταν λίγο πιο ειλικρινείς για την πολιτική που έχουν ή για το ότι δεν έχουν πολιτική. Δεν θα ήταν πιο σοβαρό να πούνε ότι, κοιτάξτε, ε, αυτή είναι η αμερικανική μέθοδος, είμαστε σκληροί και κάνουμε ό,τι μας έρχεται. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Ας πούν αυτό, είμαστε σκληροί, είμαστε μεγάλη χώρα, είμαστε ισχυρή χώρα. Ε, καλά, τότε θα λέγαμε πάσο. Όμως, έχουμε μπλέξει με αυτές τις κατεξοδοτησίες πράξεις. Τι να σας πω. Ελπίζω να με παρακολουθείτε, συνάδελφοι. Τι να πω, θα τα λέω όσο πιο διπλωματικά μπορώ. Αυτό όμως είναι το πρόβλημα. Και οι θυγόμενες χώρες επίσης νιώθουν έναν εξευτελισμό. Και κατακλείδει για αυτές τις χώρες και για τους πολίτες του που θίγονται. Ακριβώς πρόκειται για μεγάλη προσβολή να δέχονται τόσα όχι. Δεν έχει, έχει εξαίρεση η Ουγγαρία από το πρόβλημα αλλά άλλη χώρα δεν έχει. Οπότε αυτό δεν είναι προσβλητικό. Με τι κριτήριο γίνεται αυτό. Ακόμα και αν κανεί είναι και αυθαίρετο. Παρά είναι αυθαίρετο εν προκειμένου. Ακόμα και ένα Αμερικανό. Καλά. Ε, κατήντησα να παραμιλάω, αλλά τέλος πάντων. Θα πρέπει κανείς να πάει από κοντά, να επισκεφτεί το State Department, να τους δει. Τίποτα, χαμογελάνε ειρωνικά. Τέλος εντάξει, καλά καλά ξέρω ότι έχετε και άλλα θέματα που σας απασχολούν. Και τώρα, ποιος θέλει να δώσει το εκτήριο λάκτισμα. Σόφι, Μπέκερ. Όχι, είσαι κύριε Μπέκερ. So let it make me short. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Αφενός ο πρόεδρός μας θέτει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και είναι σαφές ότι οι σκέψεις του αυτές μπορούν να μας βρουν σύμφωνους. Από την άλλη μεριά δέχομαι και τις ε, σκέψεις της Επιτροπής, του Επιτρόπου και τις δικές σας για την αναζήτηση λύσεως με συνέπεια. Δεν έχω άλλο τίποτε να πω, συνεχίστε. Προσπαθήστε να επιτύχετε αυτά που σας έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Η κυρία Ιντφέλτ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα αν θα είμαστε συμπαθητικοί ή όχι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να τις υπενθυμίσουμε για ποιον δουλεύει. Και όπως σε τόσες άλλες περιπτώσεις η Κομισιόν αντιμετωπίζει ε, πολύ πιο φιλικά ή τέλο πάντων αποδίδει πολύ μεγαλύτερη σημασία στι φιλικέ σχέσει με τι ΗΠΑ από ό,τι στι σχέσει με του Ευρωπαίου πολίτε. Ο λόγο για τον οποίο δεν καταργούνται οι προξενικέ θεωρήσει για του Αμερικανού είναι. Ε, θεωρείται, θεωρώ, ε, ε, ότι να μην να μην θυγούν οι σχέσεις με τους Αμερικανούς. Αλλά για τις χώρες όπως Κύπρος, Βουλγαρία, Κροατία κλπ. Τι γίνεται. Αυτούς εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι την Αμερικανική κυβέρνηση. Και ε, είναι ακριβώ όπω σα είπε ο Κλοντ. Παίζουν παιχνίδια οι Αμερικανοί μαζί μα, Επί χρόνια. Πέρυσι είχαμε πάει εκεί το καλοκαίρι και μα είπαν ό,τι και να κάνετε δεν μα νοιάζει. Δεν θα αρθείτε ποτέ στο ύψο. Διότι σε αυτό το έγγραφό σα ένα πράγμα μόνο είναι σωστό. Όπου λέτε ότι όλο το πρόγραμμα τη κατάργηση των ψηφιακών θεωρήσεων δεν είναι σχετικό με το ταξίδια, είναι ζήτημα ασφάλεια. Αλλά να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινεί μεταξύ μα το πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων χρησιμοποιείται για να επιβληθούν αμερικανικές πολιτικές ασφάλειας στους Ευρωπαίους. Καθώς γίνεται κάποιο update, όλες οι χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Visa Waiver Program αναγκάζονται να προσαρμόζουν τις πολιτικές ασφαλείας τους. Τι γίνεται, όλοι μα θα πάμε στι εκλογέ. Μπορώ να πάω στου ψηφοφόρου μου και να πω ότι εμεί λαμβάνουμε τι δικέ μα αποφάσει εδώ στην Ευρώπη. Όχι. Διότι οι Αμερικανοί αποφασίζουν και του υποστηρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να ντρέπεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα χάλια τη. Και το ίδιο και το Κοινοβούλιο. Διότι εμείς εδώ είπαμε, είπε δηλαδή η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ότι θα πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ εκεί σταμάτησε την προσπάθεια αυτή η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Σταματήστε να παίζετε με τα παιχνίδια. Α, συζητούμε του Αμερικανού, παρακολουθούμε την κατάσταση, βοηθούμε τι πέντε χώρε. Ξέρετε, κυρία Μίχου, και ξέρει και ο Επίτροπο, γνωρίζει πολύ καλά ότι Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να διασφαλίσει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη θα συμμετέχουν στο Visa Waiver Program. Το ξέρετε πολύ καλά και μας θεωρείτε ανόητες εμάς εδώ. Και το άλλο θέμα είναι, πρόκειται για ζήτημα αρχής. Δεν είναι ζήτημα ε, ποσοστών απορρίψεων αιτήσεων για προξενικές θεωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε αρνούνται να αναγνωρίσουν τι δικέ μα εδώ θεσμικέ ρυθμίσει. και για αυτέ τι περίφημε διατλαντικές σχέσει που σα φαίνονται τόσο πολύτιμε και πρέπει θα πάμε να φιλούμε τα πόδια των Αμερικανών διότι αλλιώ δεν θα μα αγαπούν ίσως να έχετε, να έχετε λάβει υπόσχεση σα ότι μείωσαν το διπλωματικό καθεστώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί καν να μα το κοινοποιήσουν. Γιατί λοιπόν πέφτουμε στα τέσσερα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το ίδιο κι εμείς. Ε, τι γίνεται, ποιοι είναι οι συνομιλητές μας, η κυβέρνηση του Τραμπ δεν μιλούν τη γλώσσα της διπλωματίας και των σχέσεων. Ο μόνος τρόπος για να τους αναγκάσουμε να καταλάβουν είναι να τους δείξουμε ποιες είναι οι συνέπειες. Πότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ευθύνες της. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να προσκαλούμε ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσα χρόνια μας λένε τα ίδια πράγματα. Α, μιλούμε με τους Αμερικανούς, συνομιλούμε με Μα σας παρακαλώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσέλθει ξανά εδώ όταν θα έχει επιτύχει αποτελέσματα. Πρόεδρος. Εγώ πάντως ευχαριστώ την κυρία Μίχου που έκανε τον κόπο να προσέλθει ενώ γνωρίζει ότι είναι ευαίσθητο το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήλθατε και ποτέ δεν θα ήθελα να είμαι δυσάρεστος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι περίπλοκο το καθήκον σας και εσάς και σας δυσκολεύουν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, από αυτά που είπε η Σοφία, αλλά και ο κ. Μπέκερ, να είναι σαφές για οποιονδήποτε συνάδελφο παρακολουθεί και δεν γνωρίζει καλά το θέμα. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζονται άμεσα οι προξενικές θεωρήσεις για τους Αμερικανούς υλικούς, διότι εν τέλει οι χώρες μέλη και το Κοινοβούλιο μπορούν να προβάλλουν ε, βέτο και να αυξήσουν την πίεση προς τις ΗΠΑ για τη σημερινή συνεδρίαση νομίζω πάντως για να φανεί ότι είναι χρήσιμη δηλαδή ίσως μπορούμε να σημειώσουμε ένα από τα θέματα που είπε η κυρία Ιντφέλτ ότι αν δηλαδή όντως και το λέγει και στον κύριο Μπέκερ αυτό υπάρχει το θέμα δηλαδή της ρεάλ πολιτικά το πούμε έτσι και κανείς δεν το παρανοεί δεν ναι, παρανοεί ότι άλλωστε αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό είπα και όλοι να είμαστε καλύτερα ειλικρινεί στην περιγραφή των ε, γεγονότων. Αν όντω συμβαίνει αυτό, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ασκήσει πίεση στι ΗΠΑ. Όπω λέει η Σοφή Ιντφέλτ, όταν πηγαίνουμε να δούμε το State Department μας λένε κάποιοι πολίτες είναι απειλές για την, για την ε, ασφάλεια στις ΗΠΑ... Ενώ άλλοι όπω οι Ούγγροι, α πούμε, δεν, είναι, δεν πρόκειται να έρθουν εδώ στι ΗΠΑ με προξενική θεώρηση και μετά να εξαφανιστούν κάπου. Όταν λένε λοιπόν τέτοια πράγματα και μετά ταυτόχρονα. Δεν δέχονται καν τον πρέσβη μας που είναι από τα χειρότερα πράγματα. Ενώ ο νέος Αμερικανός πρέσβης είναι συμπαθέστατος. όντω ασκούν ένα είδο real Το θέμα είναι όμω ουσιώδε. Και διορωτώ με, εάν Ίσως όντως για κάτι τόσο ουσιαστικό όπου υπάρχει μια αυθαίρετη κρίση σε βάρος ορισμένων χωρών, μήπως πρέπει όντως να κάνουμε ένα βήμα. Διερωτώ με, εάν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει να αρχίζουν να πιστεύουν οι ορισμένοι ότι δεν θα είναι και ίσως αξίζει να κάνουμε ένα διάβημα, ένα βήμα προς τα εμπρός. Γιατί είναι πολύ αυθαίρετος ο τρόπος με τον οποίο διαιρούν τις ε, χώρες μέλη της Ένωσης οι Αμερικανοί. Και με κάποια κριτήρια που στερούνται λογικής. Αυτό ε, σας φαίνεται λογικό. Ε, που λέω, γιατί και αυτοί θα διαρωτώνται μέχρι πού μπορούν να το τραβήξουν, πόσο μπορούν να μας ζωρίσουν χωρίς να αντιδράσουμε. Εάν όλες αυτές οι χώρες είχαν πολίτες οι οποίοι όταν φτάνουν εκεί εξαφανίζονται, αυτό θα ήταν διαφορετική η υπόθεση. Δεν σημαίνει όμως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Ούγγροι ε, πολίτες να φτάνουν στις ΗΠΑ αντίθετα με τους Πόλωνους. Αλλά ε, να θεωρούν τους Πολωνούς ε, επικίνδυνους, αυτό είναι παράνογο. Είναι παρανοϊκό. Δεν έχει καμία ε, απολύτως βάση. Ορίστε εσείς. Για Χασάνοβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Σοφίν Τφέλτ για τα όσα είπε. Ακούμε για έκτη φορά την ίδια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία προέτους, 15 Ιανουαρίου, πέρσι. Δεν θα παραλάβω τα επιχειρήματα τα οποία ε, ανέφερε η κ. Φέλτ, αλλά έχω δύο ερωτήσεις στην κυρία Μίχου. Σε ποιο βαθμό είναι αντικειμενικά τα κριτήρια των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το 3% των θεωρήσεων που απορρίπτονται. Σε ποιες πηγές στηρίζονται σχετικά με την κατάχρηση και με την επικινδυνότητα των χωρών. Και στο ανακοινωθέν του 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να σκεφτούν ένα πρώτο βήμα, δηλαδή να κάνουν ό,τι έκανε και ο Καναδάς σχετικά με ταξιδιώτες χαμηλού ρίσκου που προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα. Στην τελευταία σας όμως ανακοίνωση δεν αναφέρεστε καν σε μια τέτοια δυνατότητα. Πότε σκέπτεστε να κάνετε τουλάχιστον αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. και μετά μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το άγχος ε, για την κυρία Μίχου. Άλλος κανείς λοιπόν. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, διότι τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Και όπως είπατε σωστά κυρία Μίχου, έχουμε άλλωστε επισκεφθεί τις ΗΠΑ Πολιτείες πολλές φορές. Βλέπετε κάποιο φως μπροστά. Και θα αλλάξουν οι διπλωματικές καταστάσεις. Βλέπετε κάποιο κίνητρο. Όχι, λοιπόν, η απάντηση σας είναι αρνητική. Να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ γνωρίζουμε πολύ καλά την απόψεις σας και ξέρετε ότι δουλεύουμε πολύ στεναρά. Ε, θα θέλαμε να μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο η ειλικρίνεια. Έχουμε νούμερα, έχουμε στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να εργαζόμαστε για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Να υπογραμμίσω το εξή ότι οι πέντε χώρες ε, που εξαιρούνται του προγράμματος απαλλαγής ε, συνεργάζονται πολύ στενά μαζί μας και ε, οι αρχές των πολιτιών έχουν προτείνει κάποιες λύσεις τις οποίες αναλύσαμε Συζητήσα, συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη και είδαμε ότι δεν είναι πραγματικές λύσεις του προβλήματος. Το η πραγματική λύση θα ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε να αλλάξουν στάση σε σχέση με αυτές τις πέντε χώρε. Εμείς εργαζόμαστε για το συμφέρον των πολιτών, όχι για τις νομες κάποια άλλη τρίτη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με βάση αυτό το κριτήριο παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Τώρα, για το, το ερώτημα το οποίο μετέθη, για την έκθεση του 2016, για τους ταξιδιώτες μικρού χαμηλού κινδύνου και την υπόθεση του Καναδά και θα επανέλθω στον Καναδά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε παρόλο που δεν αναφέρεται στην έκθεση είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό παρανομαστή, μια λύση για τον Καναδά. Για τον Καναδά, και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, πριν από μερικούς μήνες είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Καναδάς ήθελε θέλησε να απαγορεύσει την είσοδο στους Ρουμάνους πολίτες γιατί το, ήταν πολύ ψηλό το ποσοστό αιτήσεων ασύλου. Και καταφέραμε να φέρουμε σε επαφή το κράτος μέλος με τις αρχές, έτσι ώστε να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και πράγματι δεν συνέβη. Άλλαξε η στάση του Καναδά. Δεν λύνονται πάνω τα προβλήματα κάνοντας θόρυβο και οχλαγωγώντας. Προσπαθούμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους για να λύνουμε τα προβλήματα. Και τα πέντε κρατημέλη στηρίζουν την στάση μας. Γνωρίζω την θέση σας, Πρόεδρε. Δεν μπορώ βέβαια να σας δώσω κάποια υποχρέωση, ε, υπόσχεση επουλάς Κομισιόν. Ε, η ανακοίνωση δεσμεύει την κομισιόν γιατί η κομισιόν είναι ένα συλλογικό όργανο. Όμως σας εγγυώμαι. Σας διαβεβαιώνω ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Θα επανέλθουμε, αλλά ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κάποιες πρακτικές λύσεις. Έτσι ώστε για κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη τουλάχιστον να λυθεί το πρόβλημα με τον τρόπο τον οποίο επιθυμούμε όλοι. Πρόεδρος. Για να μην ότι εγώ τρελάθηκα, ε, να πω το εξή. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό που έκανε ο Καναδάς αλλά κανείς δεν λέει ότι δεν είναι δικαίωμά τους αν αυτό πιστεύουν για τη Ρουμανία. Αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι είναι κάτι διαφορετικό. Λένε δεν υπάρχει πρόβλημα με τη Σλοβακία, δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ουγγαρία, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη Γαλλία, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την Πολωνία και ένα τεράστιο πρόβλημα με τη Ρουμανία. Και δεν εξετάζουν καν τα ποσοστά απόρριψη. Ε, παίρνουν αυθαίρετες αποφάσεις. Κανείς δεν αμφισβητεί τους βασικούς κανόνες. Αυτό που έκανε ο, ο, ο Καναδάς δεν ήταν σωστό, αλλά ήταν κυριαρχικό του δικαίωμα. Ήταν κυριαρχικό δικαίωμα να άρει τη διευκόλυνση αυτή που είχε παράσει στη Ρουμανία. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις αυτές. Εδώ οι Ηνωμένε Πολιτείε δρούν αυθαίρετα, διότι δεν βασίζονται σε τίποτα. Ζητήσαμε τα νούμερα από το Υπουργείο Εξωτερικών και ήταν σαφές ότι δεν βασίστηκαν σε αυτά τα στοιχεία για την αποφασή του Ήδη το παραδέχτηκαν αυτό. Και δεν έχουν κάνει την αξιοπρέπεια να χρησιμοποιήσουν σωστά τα νούμερα. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται εκεί μέσα στον κατάλογο των πέντε, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούν και εκεί. Και αυτέ. Και ποιο ξέρει ποιε άλλε χώρε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια είναι τα ποσοστά <laughs> για την Ιρλανδία και α αφήσουμε εκτό το Ηνωμένο Βασίλειο, για την Ιρλανδία και άλλε χώρε τη Δυτική Ευρώπη. σοφή. Η κυρία Ιντβέλτ. Να καταγραφεί παρακαλώ ότι η Κομισιόν δεν απάντησε σε κανένα από τα επιχειρηματά μας, απλώς επαναλαμβάνει την ίδια άποψη. Δεύτερον, το χειρίζεστε συνεχώς σαν να πρόκειται για διμερές θέμα μεταξύ ενός κράτους μέλους και των ΗΠΑ. Όχι, πρόκειται για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Πώς είναι το ένας Πολωνός, ένας Κροάτης, ένας Βουλγάρος, Βούλγαρος πολίτης να είναι κίνδυνος, να είναι απειλή. Αν όλοι οι Αμερικανοί πολίτες είναι ίσοι ενώπιον στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν σημαίνει το ίδιο και από την πλευρά των ΗΠΑ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ε, θα συνεχίσετε την ίδια άγουσα, χωρίς να ακούτε καθόλου τα επιχειρήματά μας. Και αυτή η άγουσα δεν μας έχει οδηγήσει πουθενά μέχρι τώρα. Ναι, ναι, Όσον αφορά την Αμερικανική Κυβέρνηση Επιτροπή, τώρα έχουμε τη δεύτερη ε, ανακοίνωση όσον αφορά πάλι την ε, αναστολή της ε, απαλλαγής υποχρέωσης. Η κυρία Μίχου. Αυτή είναι η δεύτερη σχετική έκθεση, η οποία και αυτή εγκρίθηκε στις 19 12 Θεωρήσαμε ότι όλες οι αξιολογηθήσεις χώρες Τρεις τη Λιγκτονία, πέντε Δυτικά Βαλκάνια συνεχίζουν και πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή. Επίσης, Και έχουμε ένα έγγραφο εργασία, εκεί έχουμε όλα τα σχετικά στοιχεία. Δελεγώς όλε αυτέ οι χώρε έχουν αναλάβει πρωτοβουλίε και αυτά όλα τα οποία είχαμε επισημάνει στην πρώτη έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό απαλλαγή από την υποχρέωση και ακολούθησαν όλε μα τι ε, συστάσει. Όμω θα πρέπει οι μεταρρυθμίσει να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να πιάσουν τόπο και έτσι να μην ε, έχουμε πίσω γυρίσματα σε σχέση με αυτά που έχουν πετύχει τώρα όσον αφορά τα της νόμιμης μετανάστευση, τα σχετικά προβλήματα. Οι χώρες αυτές συνεχίζουν να θεσπίζουν κάποια μέτρα ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την παράνομη μετανάστευση. Επίσης έχουμε δει τι γίνεται όσον αφορά την άρνηση ε, και επίσης ε, τις αιτήσει ε, παροχής ασύλου από Ουκρανία, Γεωργία, Μολδοβία και σε σχέση με την Αλβανία το 2018 είδαμε να επιδρώνεται κάπως η κατάσταση αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τα πράγματα τώρα ξανά είναι σε καλό δρόμο και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση και ούτως ώστε να αξιοποιηθούν και να συνεχιστούν οι καλέ επιδόσει. Επίση, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για τι χώρε που δεν χρειάζονται βίζα, ούτω ώστε να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική θεωρήσεων τη ε, Ένωση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερω για την Σερβία και τα λέμε στην έκθεση. Έκανε ό,τι ζητήσαμε. Η Σερβία κατήργησε ε, την ελεύθερη διακίνηση με το Ιράν τον Οκτώβριο του 2018 Διαπιστώσαμε ευθύ αμέσω τη συνέπεια όσον αφορά την κατάχρηση στα παραθυράκια του συστήματος όλα αυτά. Συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή εύρεθμα για όλες τις Δυτικών Βαλκανίων και Ανατολικής ε, γειτονίας. Γενικά είναι πολύ καλές οι επιδόσεις όσον αφορά του ε, τους Και θα υπάρξει υποστήριξη προς αυτές τις χώρες για τη διαχείριση ε, της ε, λάθρου μετανάστευσης. Βέβαια αυτοί έχουν την κυρία Σορμοδιώτα και η Ελβανία η πρώτη είναι που υπέγραψε τη συμφωνία. 15 Ιανουαρίου, Έχω στο πρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνία με ε, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη έχουν μονογραφεί και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο που έχουν ολοκληρωθεί θα οδηγήσουν σύντομα εις την μονογραφή της συμφωνίας τώρα. Για το οργανωμένο έγκλημα και τη δημοσία τάξη όλες οι χώρες αναφέρουμε ότι συνεχίζουν τη λήψη μέτρων, ούτως ώστε να υπάρξει πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά χρειάζεται να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες. Παρά κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση του εγκλήματος θα πρέπει να γίνουν σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και άλλες προσπάθειες για διαφθορά. Χρειάζεται να κάποια μέτρα σε Ουκρανία, Μολδαβία, και κατακρίτη πρέπει να σας πω ότι η υλοποίηση των κριτηρίων για την εξαίρεση της βίζας είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται και θα χρειαστεί περαιτέρω ε, εποπτεία. Οπότε προσπαθούμε από Επιτροπής στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία να έχουμε σύντονες προσπάθειες να ελέγχεται η κατάσταση και στις προσπαθίες μας για πρόοδο ξέρουμε ότι στο πλάι μας και το Κοινοβούλιο Χρυσή η θέλει το λόγο. Ευχαριστούμε κυρία Μίχο για την πλήρη εκθεσή σας, πρώτη και την δεύτερη όσον αφορά το μηχανισμό αναστολή της απαλλαγής για τη θεώρηση και κάπως όμως εξεπλάγει όσον αφορά τον μηχανισμό αναστολής ο οποίος προβλέπεται ούτω ώστε να είναι κάποιο είδου εξασφάλιση όσον αφορά την απαλλαγή της υποχρέωσης. Όταν έγινε αυτή η απαλλαγή για τις βαλκανικές χώρες, είδατε, ή μάλλον μας είπανε πολλοί, ότι έχουμε κάποιες ροές μεταναστευτικές από τα Βαλκάνια που θα μπουν με την απαλλαγή της θεώρησης στην ε, Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει όμως τώρα. Έχουμε νόμιμη μετανάστευση. Αλλά που δεν όμως αναφέρεται στο κείμενό σας. Είναι δύσκολο να καταλάβω τελικά τι ισχύει για τον μηχανισμό όταν θίγεται μόνο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Τι θα γίνει, θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα σκιάχτρα, τους μύθους για την μετανάστευση. Δεν θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη των νομίμων ροών. Αυτό ισχύει επίση και για τις χώρες της Ανατολικής ε, Και ακόμα περισσότερο. Γιατί λαμβάνοντα υπόψη σχετικά αριθμητικά στοιχεία για την ε, νόμιμη μετανάστευση από πλευράς ε, Ανατολικής Γετνίας, ε, βλέπουμε ότι είναι εντυπωσιακά κάποια από αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Η Ουκρανία ε, είναι οι πρώτοι που θα οφειλθούν από την άδεια ε, διαμονή στην Ένωση. Το 17 βλέπουμε ότι έχουμε Έχουν περίπου 660.000 περίπου. Και στη Γαλλία είπαν ότι πρόκειται για βοήθεια προς την Ευρώπη όσον αφορά την κρίση. Αλλά αυτοί δεν είναι πρόσφυγες. Αυτές οι άδειες που δίνονται 85% στην Πολωνία είναι άδειε διαμονή για λόγους οικονομικούς. Και έχουμε όλο ένα περισσότερες τέλο πάντων τέτοιες άδειες. Αλλά ακριβώς και μόνο αυτού του μηχανισμού μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας που είναι το 20% του συνόλου. Να, πώς προκύπτει η αύξηση της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν είναι από νόμιμους ετούντες ε, άσυλο. Δεν δίνονται σε αυτούς ε, ε, οι άδειε διαμονής για λόγους διεθνούς προστασίας. Άρα θα πρέπει στο θέμα του μηχανισμού να λέμε και για την νόμιμη μετανάστευση και να μην εξετάζουμε μόνο τη λαθρομετανάστευση. Άλλιως δεν έχουμε συνολική εικόνα. Όχι, δεν έχω τίποτα με την ε, Πολωνία. Με ενδιαφέρει το Ουκρανικό. Όμως θέλω να ισχύουν τα ίδια πράγματα για όλους. Είδατε όμως τι λέει για την νόμιμη μετανάστευση, για την οικονομική μετανάστευση η Πολωνία και από την άλλη μεριά για το θέμα της διεθνούς προστασίας. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να έχουμε τη συνολική εικόνα για το θέμα. Καλά, λέει ο Πρόεδρος. Δεν θέλει άλλο το λόγο. Ωραία, τότε για κυρία Μίχου, τελευταία παράκληση να μας απαντήσει. Όπως σωστά είπατε, αυτή η έκθεση εστιάζεται πιο πολύ στα benchmarks, ε, στα συγκριτικά κριτήρια τα οποία έχουμε καθορίσει. Καταλαβαίνω την άποψή σας, τη σημειώνω. Να σας πω όμως ότι συζητήσαμε και με τα κράτη-μέλη και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους οι χώρε τη ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Καταλαβαίνω βέβαια ότι χρειάζεται περισσότερες πληροφορίε γι' αυτό. Πάντως, οι διμερείς σχέσεις είναι σημαντικές, ε, αλλά δεν πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται σε τέτοιου Ευχαριστώ πολύ κυρία Μίχου. Ξέρουμε ότι έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αντιλαμβανόμαστε και εσείς ότι τα θέματα αυτά έρχονται και ξανάρχονται και ξαν... κάθε φορά ε, απευθυνόμαστε στην Κομισιόν για απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω τον ομιλητή, μιλάει χωρίς μικρόφωνο. Ναι, thank you. What, what is it about you, Juan? Τι έχεις εσύ με την κυρία Μίχο ακριβώς. Ε, άκουσα τι είπες, αλλά Πώς τη γοητεύεις τώρα την κυρία Μίχου τόσο πολύ. Ε, σε ζηλεύω. Είπε ότι πρέπει να φύγει και εσύ τη ζήτησες τώρα να μείνει και είπε με χαρά δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει μεταξύ σας. Ωραία. Θα μείνει η Κομισιόν για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα για τις θεωρήσεις που εισηγητή είναι ο κ. Αγγιλάρ. Τι έγινε μετά το δεύτερο τριμερή διάλογο. Παρουσία της κυρίας Μίχου. Θα είμαι σύντομος. Γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Είναι ένα νομοθετικό θέμα αυτό, είναι νομοθετικό ε, ζήτημα, αφορά τον κώδικα για τις θεωρήσεις, ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν από την αρχή της θητείας της ε, κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου. Όταν αντιμετωπίζαμε σημαντικά προβλήματα, ε, έχει έρθει η ώρα να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε με τη βοήθεια της Κομισιόν και ελπίζουμε με κάποιους συμβασμούς από πλευρά του Συμβουλίου. Να σας αναφέρω που βρίσκεται η κατάσταση στο θέμα των τριμερών διαλόγων. Τελευταίος έλαβε χώρα το Δεκέμβρη, 17 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, στο Στρασβούργο, με την ευκαιρία της τελευταίας ολομέλειας του χρόνου. Από τότε και μετά έχουν λάβει χώρα και συναντήσεις με τους ε, μεταξύ σχεδόν συγκριτών και συγκριτή και τεχνικές ε, συναντήσεις και η θέσπιση αυτού του κώδικα θεωρήσεων απαιτεί να βιαστούμε έτσι ώστε στις 29 Ιανουαρίου στον επόμενο τριμερή διάλογο που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το ζήτημα είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε συμφωνία του Κορεπέρ το Φεβρουάριο και, η, και ψηφοφορία στη Λίμπε 18-19 Φεβρουαρίου έτσι ώστε να ψηφιστεί στην δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να αποφύγουμε κόκκινες γραμμές κατά το δυνατόν και να κάνουμε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς για τα εκκρεμή θέματα. Όπως θυμάστε, συζητούσαμε το θέμα της συνεργασίας για την ε, διάταξη βανισδοχής, ενδέεται με το άρθρο 25. Συμφωνία αντιπροσώπευσης βρήκε αντίθετα, αντίθετα πολλά κρατημέλη, ορισμένα από τα μεγάλα μάλιστα. Επίσης, συζητεί το θέμα των προθεσμιών του άρθρου 9 για τις, ε, την ε, υποβολή ετοιμάτων, ε, το θέμα της ιατρικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια ταξιδιών. Δεν υπάρχει, υπάρχουν στοιχείο που να απαιτούν την ύπαρξη τέτοια ασφάλεια, οπότε θα πρέπει να διαγραφεί κατά άποψή μα. Μετά έχουμε τις, τα τέλη για την έκδοση θεωρήσεων και των συναφών υπηρεσιών. Τα άρθρα 1, 2 και 16 που αναφέρονται στους ε, επαγγελματίες του πολιτισμού και του αθλητισμού θα πρέπει να διευκολυνθούν και προθεσμία για να ληφθεί η απόφαση του άρθρου 23. Επίσης συζητήσαμε τις ε, θεωρίες πολλαπλής εισόδου ε, για το... Ε, για, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ε, πολλαπλή είσοδος και έξοδος. Και επίσης συζητήσαμε το θέμα της χορήγησης θεωρήσεων στα εξωτερικά σύνορα υπό προϋποθέσεις. Έχουμε πολλούς συναδέλφους εδώ που ήταν σκιοδησηγητές και στο παρελθόν και ξέρουν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να είναι απόλυτα ξεκάθαρο το κείμενο και να συμφωνήσουμε, να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό έγκαιρα. Νομίζω ότι αυτός ο κώδικας θεωρήσεων θα μπει στο κομμάτι του, ε, των πολύ θετικών νομοθετικών κειμένων που θα έχουμε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ζητώ από τους διερμηνείς να συνεχίσουμε μερικά λεπτά. Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε δύο-τρία άτομα που ουσιαστικά που θέλουν το λόγο να τους ακούσουμε. Ποιος Μπέκερ από το ΕΛ καταρχήν. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τη γενική τοποθέτηση του εισηγητού. Θεωρώ εκτιμώ μάλλον πολύ θετικά την ρεαλιστική προσέγγιση του εισηγητού σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και ταυτόχρονα Χαίρομαι για τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο και τα τρία μέρη, μεταξύ αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητούν συμβιβασμό. Δεν θα σας κρύψω ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες θέσεις όπου εγώ αισθάνομαι κοντά σε Επιτροπή και Συμβούλιο. Συμφωνώ όμως ε, με τη γραμμή που προτείνει ο εισηγητής μας και ελπίζω ότι θα αποβεί επιτυχής. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούμε και ευχαριστώ εσάς προσωπικά κυρία Μίχου, διότι είστε των διαπραγματεύσεων από πλευρά Κομισιόν και εκτιμώ πολύ και την προσωπική σας ε, στράτευση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ... Ε, και εγώ βεβαίως, ε, πολύ σωστό αυτό που λέτε, και εγώ βεβαίως ευχαριστώ την κυρία Μίχου για όλη την προσπάθεια ε, στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πέκερ. Ναι. Ο κ. Ντεπρέ ω σκιώδης ε, των ε, φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Σημαντικό το το οποίο ε, ξεκίνησε με αρκετό κόπο, αλλά τώρα έχει πάρει φόρα. Η πολιτική μου ομάδα θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγκριθεί ήδη εντό τη παρούσα κοινοβουλευτική θητεία το θέμα. Αντίθετα με τον κύριο Μπέκερ, η δική μας ε, ομάδα προσεγγίζει περισσότερο στην θέση του ε, Κοινοβουλίου και όχι του Συμβουλίου. Τονίζω τώρα δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, χαίρο γιατί για το ευαίσθητο θέμα της πολιτικής θεωρήσεων και για να ενθαρρυνθεί η ε, σχέση με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή, ο εισηγητής μας μπόρεσε να πει στο Συμβούλιο να διαπραγματευτεί στη βάση των προτάσεων του Κοινοβουλίου. Διότι εμείς δεν θέλαμε ε, ο πληθυσμός των ε, χωρών αυτών ε, να υφίσταται τις συνέπειες της έλλειψης συμφωνίας επανεισδοχής με την Ευρώπη. Και μάλιστα το τέλο για την προξενική θεώρηση περνά από 80 ευρώ στο διπλάσιο, το οποίο για ορισμένου από του ανθρώπου αυτού είναι απαγορευτικό. Θα ήθελα λοιπόν να προβλεφθεί μια πολιτική η οποία να δίνει και κάποια θετικά ε, κίνητρα, μειώνοντα α πούμε το ε, το κόστο των θεωρήσεων για του ε, πολίτε των χωρών εκείνων οι οποίε συνεργάζονται σωστά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιρήτα. Τώρα έχουμε ακόμα πολλή δουλειά με το φάκελο αυτό. Η συμμετοχή των χωρών μελών. Οι ε, θεωρήσεις για καλλιτέχνες που βρίσκονται σε τουρνέ και ούτω καθεξής. Εγώ πάντως εμπιστεύομαι τον εισηγητή μας, τον υποστηρίζουμε για να προλάβουμε και τις προθεσμίες που έχουμε όλοι μαζί εγκρίνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ζεράρ. Θα μας εγκαταλείψουν τόσο λίγο οι διερμηνείς. Παρακαλώ Μαρή Κριστίν σύντομα. Δεν θα καταχραστώ ούτε του χρόνου των ε, διερμηνέων ούτε του χρόνου της κυρίας Μίχου. Δεν θα επανέλθω στο ιστορικό του φακέλου που είναι όντως περίπλοκο. Θα επιμείνω σε ένα θέμα που μου φαίνεται σημαντικό. Διαφωνώ σε ορισμένα σημεία. Αλλά ε, ας πούμε, ας δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά. Ο Ντεπρέ μίλησε για την επανεισδοχή και συμφωνώ με αυτό που είπε. Επιμένω σε τρία θέματα. Πρώτον, η ιατρική ασφάλιση. Δεν θα πω περισσότερα. Τουρνέ καλλιτεχνών και αθλητών. Ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε πάρα πολύ συχνά και πολλές παράπονα, παράπονα και καταγγελίες και πραγματικά εκεί υπάρχει μια σύγχυση. Και τέλος, θεωρήσεις στα σύνορα, εμένοντας το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει σήμερα. Και δεν κατανοούμε για ποιο λόγο πάνε να την καταργήσουν διότι είμαι βεβαία ότι οι χώρες οι οποίες είναι ε, όμορες χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις που πρέπει να τις ρυθμίζουν στα σύνορα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη δυνατότητα να χορηγούνται οι θεωρήσεις ε, στα σύνορα. Αλλιώ πρόκειται για υποχώρηση η οποία θα ζημιώσει του πάντε. Ευχαριστώ, Μαρία Κριστίν. Ευχαριστώ που υπήρξε σύντομη. Κύριε Μίχο, εσεί ε, ηγείστε των διαπραγματεύσεων και του τελευταίου τριμερού διαλόγου. Έχετε να πείτε δύο λόγια. Πολύ σύντομα. Συμμετείχα στον τριμερή διάλογο, κάτι το οποίο θεωρώ τιμή μου και προσπαθήσαμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εξέβρεση μιας λύσης θα είμαι και στον επόμενο τριμερή διάλογο και ο ίδιος επίτροπος θα είναι μάλιστα. Άρα, από τώρα μέχρι τον τριμερή διάλογο θα πρέπει να κάνουμε πάντα δυνατόν για να βρούμε λύσεις. Για να μπορέσει να γίνει ο τελευταίος τριμερής διάλογος. Τα ζητήματα που τονίσατε κι εσείς είναι αυτά που συζητούνται. Δεν μπορώ να σας πω ότι όλα όσα είπατε θα συζητηθούν στον, τελευταίο τριμερή διάλογο για διαφόρους λόγους αλλά προσπαθούμε να παραμείνουμε ως το δυνατόν εγκύτερα στις... Ναι, όσο το δυνατόν εγκύτερα, επαναλαμβάνω, στα όσα είπε ο εισηγητής σας, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα επιδέξιος και βοηθεί ώστε να ε, συμβάλλουμε όλοι προς την διακατεύθυνση. Ευχαριστώ και τους τρεις, ευχαριστώ κυρία Μίχου. Βλέπω ότι είστε επιδέξιος και στις γλώσσες. Α, σε μεγάλη φόρμα σήμερα, ε, Χουάν. Ευχαριστώ κύριε Μίχου. Ε, πρόεδρος, ευχαριστεί και όλα τα μέλη και βεβαίω ήμουν και εγώ στον τριμή διάλογο της Δευτέρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ωραία τελειώσαμε τη συνεδρίαση. colleagues, next meeting is... Και η επόμενη συνάντησή μας 29 Ιανουαρίου. Πέρα τη συνεδρία σα. Ευχαριστούμε και του διερμηνεί. Nice την παράταση που έδωσα.